Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας αρχίσουμε, ας ε, πάψουμε τις ε, ιδιωτικές συζητήσεις και ας αρχίσουμε τη συζήτηση για τη θέση μέτρων κινητικότητας, δηλαδή να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Και το σημερινό απόγευμα έχουμε την ενιαγορά και τα σχετικά μέτρα με εισηγητές τους κυρίους Βαντεκάμπ, Κίλονεν, κυρία Κίλονεν, και την κυρία Μοντέρο που δεν είναι ακόμα παρούσα. Ας αρχίσουμε πρώτα με εσάς κύριε Βαντεκάμπ. Θα σας δώσω το λόγο. Θα ακολουθήσει η συζήτηση με τους συζήτητες και βεβαίως όπως πάντα τέλος θα ρωτήσω την γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Βαντεκάμπ, αν είστε έτοιμος, ας αρχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εδώ να μνημονεύσω τον ε, Γιάννη Νίλσον. Ήταν ένας από τους ε, τρεις ε, εισηγητές για αυτό το θέμα, για την οργάνωση της αγοράς. Έχουμε και τον φάκελο του Καμποτάς που είχε αναλάβει ο Γιέντς, της απόσπασης που είχε αναλάβει η κυρία Κίλωνεν και εγώ είμαι εισηγητής για τους χρόνους ε, οδήγησης και ανάπαυσης. Και αν ε, όντως ε, γίνει έτσι, χαίρομαι που θα αναλάβει την έκθεση του Καμποτάζ ο Ισμαήλ Ερτούκ. Όπως και να έχει κάποιος συνάδελφος από τους σοσιαλιστές. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε 294 τροπολογίες. Σημαντικός αριθμός. Και καταφέραμε να τις ε, ομαδοποιήσουμε σε νέα ενότητες, τις οποίες ε, και εξετάσαμε κατά τη διάρκεια της πρώτης ε, συνάντησης και οδών εισηγητών στις 13 Μαρτίου και την 3η 27 Μαρτίου θα γίνει η δεύτερη συνάντηση των σκιωδών και εκεί ε, θα καταθέσουμε και τις πρώτες συμβαστικές τροπολογίες. Αύριο το μεσημέρι, αν και αυτό ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει τόσο, έχουμε ήδη μια τεχνική συνεδρίαση για να εξετάσουμε μια σειρά τεχνικά ζητήματα. Οι τροπολογίες είναι πολλές, ε, έχουν διατυπωθεί με επιμέλεια και αφορούν τα εξής στοιχεία. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα της έκθεσής μου είναι η θέση των ελαφρών εμπορικών οχημάτων, των λεγόμενων LCVs. Και τις τροπολογίες ε, προκύπτει ένα αίτημα να διαβρύνουμε τον κανονισμό και για τα οχήματα κάτω από τους 3,5 τόνους. Και φτάνουμε έτσι στους 2,4, 2,5, 2,8 τόνους. Αυτό θα καθορίσει η συμβαστική τροπολογία. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή για να συμπεριλάβουμε και τα ελαφρά ε, οχήματα έχει επιπτώσεις και για τον ε, ταχογράφο αλλά και για τις προϋποθέσεις ε, θέσπισης οι οποίες θα μπουν υπό το καμποτάζ. Αλλά κατά τη γνώμη μας διαδίνονται από δύο και γίνονται τέσσερις σε τέσσερις. Μετά, Πρόεδρε, για τους χρόνους ε, οδήγησης και ανάπαυσης υπάρχουν διάφορες ε, μεταβολές σε αφορά την εφαρμογή και διάφορες, διάφοροι τρόποι εφαρμογής δηλαδή αυτής της νομοθεσίας ανάλογα με την ευελιξία που θα προβλέψουμε αλλά υπάρχουν και τροπολογίες που λένε όχι να το αφήσουμε ως έχει με βάση τον ισχύοντα κανονισμό που λειτουργεί μια χαρά στην πράξη και ε, απορρίπτουμε την ευελιξία που θέλει να προσθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα είναι ένα βασικό ζήτημα διαπραγμάτευσης λοιπόν. Ιδιαίτερη έμφαση, κυρία Πρόεδρε, ε, δίδεται στις ε, μεταφορές μέσω λεωφορείων. Κάποιοι θέλουν να βάλουμε στο ίδιο καζάνι τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Αυτό κατά τη γνώμη είναι αντιπαραγωγικό, ιδίω για του οδηγού λεωφορείων. Εάν ένα οδηγό λεωφορείο έχει ένα λεωφορείο με 50 επιβάτε, είτε αυτό είναι για μικρή είτε για μεγάλη απόσταση, αυτό ε, προποθέτει διαφορετικό καθεστώ ανάπαυση από ότι σε ένα ε, φορτηγό. Πρέπει να εξετάσουμε τον κανόνα των 12 ημερών, να το διευρύνουμε και σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν τροπολογίες για την ημερήσια ανάπαυση. αλλά και άλλες τροπολογίες για τη διατήρηση της ε, σύντομης ανάπαυσης. Τέταρτη ενότητα. Συσσωρευμένος χρόνος οδήγησης. Ορισμένοι συνάδελφοι και από το ΕΛΚ έχουν καταθέσει τροπολογίες σε ό,τι αφορά ε, το σύνολο των ε, ορών εργασίας και θα, θα διαβριθεί κατά τη γνώμη τους στις 180 ε, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα το συζητήσουμε περαιτέρω για να καταλήξουμε σε συμβαστική τροπολογία. Πέμπτο σημείο. Είναι ε, η ε, ανάπαυση μέσα στην ε, καμπίνα οδήγηση. Σε ορισμένε χώρε όπω η Γερμανία και η Γαλλία αυτό απαγορεύεται, ιδίω σε ό,τι αφορά την εβδομαδιαία ανάπαυση αλλά σε άλλες χώρες είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η ευελιξία της ανάπαυσης στην καμπίνα. Και όπως είδατε προτείνω να συνδυαστεί αυτή η ανάπαυση στην καμπίνα με ασφαλείς ε, χώρους στάθμευσης. Αυτός ο συνδυασμός θα τεθεί υπό συζήτηση βέβαια γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε συμβασμό. Επόμενο σημείο, η επιστροφή στην έδρα. Πότε επιστρέφει κανείς στο σπίτι του, μετά από τρεις εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες. Επιστρέφεις στη σύζυγο ή στη φίλη σου ή και στις δύο. Ολόκληρη συζήτηση ήταν και αυτή. Αλλά πρέπει και πάλι να προσέξουμε. να μην ακολουθείς μια πεταναλιστική προσέγγιση. Και αυτό το επιστροφή στο σπίτι ίσως θα πρέπει να το, να το αντικαταστήσουμε από μια άλλη καλύτερη διατύπωση, έναν κατάλληλο χώρο ανάπαυσης. Και βέβαια το ερώτημα είναι ποιος θα το πληρώσει όλο αυτό. Ξέρω ότι σας δυσκολεύει η έννοια σύντροφος, φίλη, αλλά πρέπει να το συνηθίσετε, γιατί το ΕΛΚ είναι πολύ μοντέρνο κόμμα. Το πρώτο τελευταίο, η επιβολή του νόμου. Πολλοί από αυτούς ε, τους χρόνους ε, ανάπαυσης και σχετικές νομοθετικές διατάξεις απλώς ε, δεν εφαρμόζονται από, την, από τα Γιατί δεν έχουν τη χρηματοδότηση, δεν θέλουν να, να δαπανίσουν αυτά τα κονδύλια, ούτε τον εξοπλισμό για να έχουν ταχογράφους και βέβαια πολύ περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουν υποβληθεί λοιπόν πολλές τροπολογίε σε αυτό το σημείο. Προς το παρόν υπάρχει ένα σύστημα, το ERRU, και θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το διευρύνουμε ή να το βελτιώσουμε. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα ούτε για τους εργαζόμενους, να εξετάσουμε το θέμα των χρόνων οδήγηση και ανάπαυση, εάν δεν εφαρμόζονται τελικά οι κανόνε. Και αυτό είναι και μια προειδοποίηση προ το Συμβούλιο, γιατί εμεί μπορούμε να σα ε, φτιάξουμε την καλύτερη νομοθεσία και να ε, συμφωνήσουμε. Αλλά αν τελικά τα κράτη-μέλη δεν την εφαρμόζουν, τότε όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Κλείνοντα, Πρόεδρε, ο διαβόητο ταχογράφο. Προτείναμε ε, να εισαγάγουμε τον FEE ταχογράφο στην 1 την 1η Ιανουαρίου 2020. Πολλές τροπολογίες στηρίζουν αυτή την πρόταση, κάποιες ε, κάπως την αναβάλουν. Και εδώ θα πρέπει ε, να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να πεθύνω ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία την περασμένη εβδομάδα ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με προβλήματα για το type approval και τις απαιτούμενες λειτουργικότητας σε ό,τι αφορά την καταχώρηση, τη διασυνοριακή καταχώρηση. Ε, Πολύ καλά έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημέρωσε το Συμβούλιο, αλλά θα ενημερώσει και το Κοινοβούλιο ή εμείς είμαστε αμεληταία ποσότητα και δεν την ενδιαφέρει να μας ενημερώσει. Ε, θέτω απευθεία το ερώτημα για να ξέρουμε κι εμείς που βρισκόμαστε. Αυτά εν είδη εισαγωγής, κυρία Πρόεδρε. Στον φάκελο για το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βαντερκάμπ. Ας ε, ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση. Η Ζέμερλα Δερμόντε για τους σοσιαλιστές. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, όχι μόνο για τη δουλειά του, αλλά για την συμμετοχή που, όπως είπε, είχαμε πολλές καρπαφόρες συναντήσεις των σχεδόν. Πρέπει όμως να, συμφωνήσουμε και για τις άλλες εκθέσεις που σχετίζονται με αυτό το θέμα, ώστε να υιοθετηθεί το πακέτο αυτό μέχρι το τέλος της θητείας. Μετά μου φαίνεται φυσιολογικό να υπάρχουν βέβαια διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά είναι απαραίτητο νομίζω να βρούμε μια σύγκληση σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα, βιωσιμότητα των μεταφορέων, και τη δημιουργία μια πραγματικά ανταγωνιστική ενιαία αγορά που θα τηρεί κανόνες με ξεκάθαρου ελέγχους και κανόνες για όλου. Ξεκινάω με τους ταχογράφους, γιατί νομίζω ότι πρέπει εδώ κάτι να γίνει άμεσα για να έχουμε ένα έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Μετά συμφωνώ με τους εξοπλισμένους και ασφαλείς χώρους στάθμευσης για την ανάπαυση των οδηγών. Να έχουμε δηλαδή μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα ανταποκρίνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στα αιτήματα των οδηγών. Επίσης πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Μιλήσαμε για την επιστροφή στο σπίτι. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχουν παρερμηνίε. Ακριβώς για να διευκολύνουμε τους ελέγχους και να επιτρέψουμε, λέω και εγώ, στους οδηγούς να γυρίσουν στο σπίτι τους και να μην μείνουν εκτός εστίας και να καθοδηγούνται από τους επιχειρηματίες. Και κάτι τελευταίο. Μεταφορά πιβατών και λεωφορεία. Νομίζω θα πρέπει να υπάρξει χωριστή νομοθετική διάταξη γι' αυτό. Γιατί υπάρχει διαφορά. Είναι τελείως διαφορετικό έδος μεταφοράς αυτό. Οπότε θα πρέπει να βρούμε κάποια διαφορετική νομοθετική λύση. Εμείς θεωρούμε θα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση διαφορετική όσον αφορά τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, τηρώντας πάντα βέβαια τα κοινωνικά δικαιώματα των οδηγών και προ όφελο τη ασφάλεια. Αλλά θα πρέπει βέβαια να επιδείξουμε και κάποιε ευελιξίες. Καταλήγω λέγοντας ότι παραμένουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα τα οποία όμως νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε στις επόμενες συναντήσεις του σχεδόν. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Ντεμόντε. Σεις κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα τον Βιμ Βαντεκάμπ. Τώρα μας λείπει τόσο ο Νίλσον, ο συνάδελφός μου που αποβίωσε τόσο ξαφνικά και βεβαίως τον σκεπτόμαστε διαρκώς. Βλέπουμε και το όνομά του στην ημερήσια διάταξη. Τώρα, για, τις, ε, για τους χρόνους αναπαύσεως. Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα μια συνάντηση των εισηγητών. Καλά τα πάμε στη συνεργασία. Συμφωνήσαμε στην αρχή σε πολλά πράγματα. Τώρα βέβαια σιγά σιγά αρχίζουν και φαίνονται και οι διαφορές απόψεων. Σημαντικό πάντως είναι να δούμε ότι οι χρόνοι αναπαύσεως έχουν αποδείξει την αξία τους και να δούμε τώρα πώς θα τους ρυθμίσουμε. Έχω ορισμένα πράγματα τα οποία ήδη συζητήσαμε και που κατά την άποψή μου είναι σημαντικά. Αφενός τα ελαφρά οχήματα ελαφρά φορτηγά οχήματα. Δεν πρόκειται μόνο για την κλάση βάρους. Καθώς και αν θα ισχύουν αυτά τα πράγματα εθνικά ή και διεθνώς. Μπορεί να υπάρχει για παράδειγμα αυτοκινήτο το οποίο κάνει διαμεθοριακά παραδόσεις ψωμιού. Επομένως δεν μπορεί να αποκλείεται μια ρύθμιση για να ισχύσει διεθνώς εφόσον ισχύει στο εθνικό επίπεδο πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πρακτικές, ρεαλιστικές λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις. Εξάλλου, ο ορισμός του τι σημαίνει home, δηλαδή στο σπίτι του, να γυρνάει κάποιος στο σπίτι του. Βεβαίως θα πρέπει ο οδηγός να μπορεί τακτικά να περνά χρόνο στο σπίτι του. Δεν μπορεί όμως να εξαναγκαστεί να πάει σπίτι του εάν για κάποιο λόγο δεν θέλει. Είναι βέβαια δύσκολο να γίνει η οριοθέτηση και πώς θα το αποφύγουμε, ότι δεν μπορούμε σε κάποιον να δεν επιτρέπεται να πάει σπίτι του. Μπορεί όμως μια εταιρεία γραμματοκιβωτή όπως λέγεται, δηλαδή εικονική, να μην το επιτρέπει να πάει σπίτι του. Θα πρέπει και εκεί λοιπόν να βρούμε πρακτικές λύσεις. Οδηγοί λεωφορείων και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων έχουν διαφορετικά καθήκοντα. Σωστό. Και γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη ευελιξία στις ρυθμίσεις οδηγοί λεωφορείων που φέρνουν ομάδε επισκεπτών μου, για παράδειγμα, στι Βρυξέλλε ή στο Στρασβούργο, μου λένε πάντα, κοιτάξτε, δεν έχουμε τα ίδια καθήκοντα με τον οδηγό φορτηγού. Βεβαίω και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η χρόνια αναπαύσεω και για τα πρόσωπα αυτά. Μπορεί ωστόσο οι άνθρωποι αυτοί να πάνε μία φορά σε μια κατεύθυνση και μετά να επιστρέψουν στην έδρα του και στο μεταξύ να μην οδηγήσουν καθόλου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη βέβαια και τι εξαιρέσει. Ο κανόνα είναι σαφής όμως, για τις εξαιρέσει έχω εγώ καταθέσει ορισμένες τροπολογίες. Για παράδειγμα, είχαμε προβλέψει και μια εξαίρεση για τους ε, ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα, δεν είναι όμως επαγγελματίε οδηγοί. Έχουν ταχογράφου, αλλά πρέπει αυτοί να ρυθμίζονται διαφορετικά από τον ε, επαγγελματία οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου που είναι στο τιμόνι πολλέ ώρε καθημερινά. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Νομίζω επίση θα πρέπει να είναι δυνατόν από την πλευρά των χωρών μελών να προβλεφθούν εξαιρέσει. Για παράδειγμα, για την κατασκευή οδών. Εγώ τα έχω ακούσει αυτά και για τον ταχογράφο. Εάν γίνονται έργα κατασκευή του οδού, θα πρέπει αυτό να συμπεριληφθεί ω χρόνο στο χρόνο αναπαύσεω του οδηγού. Το άλλο που μου είπαν ενδιαφερόμενα μέρη δηλαδή, εάν για παράδειγμα τον χειμώνα και σπανίζει το καύσιμο για τις θερμάνσεις, θα αφήσουν τους ανθρώπους να μην έχουν πετρέλαιο θέρμανσης μόνο και μόνο επειδή πρέπει να τηρήσουν κάποιους χρόνους αναπαύσεως. Τώρα, η ανάπαυση στην καμπίνα του ε, αυτοκινήτου. Είπαμε, κανονικά θα πρέπει να πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο για να κοιμηθούν. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε όμω καταρχήν, γιατί καμιά φορά και η θάλαμη των φορτηγών αυτοκινήτων είναι τόσο περιποιημένη που οι άνθρωποι, οι οδηγοί δηλαδή, προτιμούν να κοιμηθούν μέσα στο φορτηγό. Και τέλο ταχογράφη βεβαίω να θεσπιστεί η ρύθμιση νωρίτερα, όμω ακόμα δεν έχουμε, βεβαίως είναι όραμα του μέλλοντο η αυτόνομη ε, κίνηση των αυτοκινήτων. Αλλά κάτι να προβλέψουμε. Να μην δηλαδή εμποδίσουμε μια μελλοντική τέτοια τεχνολογική εξέλιξη. Να υπάρχουν ρυθμίσεις δηλαδή από τώρα που να επιτρέπουν την ε, κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα δηλαδή και αν ο οδηγός δεν οδηγεί καθόλου. Ευχαριστώ, έχετε δίκιο κυρία ε, Μάισνερ που λέτε ότι ήδη από σήμερα πρέπει να θεσπίσουμε πλαίσιο και βεβαίως θα κρυθεί από το αποτέλεσμα να μην τα κάνουμε έτσι ώστε να μην, να μην ε, ε, είναι δυνατόν να επιβληθεί ο νόμος όταν θα έχει εγκριθεί μέσα από τον ε, τριμμένο διάλογο. Κύριε Τέιλορ, εσείς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους άλλους συναδέλφους που μίλησαν ως τώρα. Βάντε Κάμπ, που οργάνωσε την συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Μα έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε και εμείς οι πράσινοι είχαμε την ευκαιρία να ζητήσουμε μείωση των ωραρίων οδήγηση ώστε να καταπολεμηθεί η κόπωση των οδηγών και επομένως τα συνεπαγόμενα ατυχήματα. Και με χαρά μου βλέπω ότι υπάρχει και μια διάθεση και από τα άλλα μέρη να το εξετάσουν το θέμα αυτό την Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, ακούσαμε ήδη μερικές φορές να αναφέρονται οι άλλοι, στην ευκαμψία ή ευελιξία, flexibility. Νομίζω η ευκαμψία από τη σκοπιά του εργαζόμενου δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο να οδηγούν περισσότερες ώρες ή να οδηγούν μακρύτερα από ό,τι οδηγούν τώρα. Και να, να δούμε και την διασύνδεση του καμποτάζ, της απόσπασης εργαζομένων, του, των ωραρίων οδηγήσεως και των, οδηγίων, ε, ε ωραρίων απάψεως. Στο κέντρο του κοινωνικού πυλώνα πρέπει να βρίσκεται ο οδηγός. Οδηγός ανεξαρτήτως φύλου και η κοινωνική του ή της προστασία. Απασχόλησης, σε ε, όρους θεμητού ανταγωνισμού. Να μην γίνεται dumping, κοινωνικό dumping δηλαδή, και να μην ε, ε, υπάρχει κίνδυνο να αυξηθούν τα ατυχήματα. Νομίζω τώρα και στι επόμενες συναντήσεις θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά στην ανάγκη διατήρησης της ανάπαυσης του οδηγού στο σπίτι του στο σπίτι τη η πρώην πρώτη γυναίκα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Και για να απαντήσω στον εισηγητή για το ποιο θα πληρώνει, γιατί να μην πληρώσει ο εργοδότη. Πληρώνει για την ασφάλιση ασθένεια κλπ. Γιατί να μην πληρώνει και γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι απολύτω ορθό να επιβεβαιώσουμε το δικαίωμα, τα δικαιώματα των αδειών να επιστρέψουν μεταξύ αυτών και το δικαίωμα να επιστρέψουν στην αιστεία τους. Σε ό,τι αφορά τους ευφυείς ταχογράφους, θα είναι χρήσιμος για να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νόμου. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον στόχο του 2020. Δεν βλέπω και κανένα λόγο να μην ισχύσει από τότε ο ταχογράφος, γιατί ο κλάδος μπορεί σχετικά με οικονομικό τρόπο να αναβαθμίσει τεχνολογικά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για να εξασφαλίσει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες εργασίας, εργασίας για τους οδηγούς. Και ποιος δεν θέλει αυτό να το κάνει. Η κυρία Κύλωνε, νωρίστε κυρία μου. Αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητοί και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο Βιμ για την συνεργασία, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για όλα τα θέματα. Και εμένα μου λείπει πολύ ο Γένς. Είναι ωστόσο σημαντικό να συνεχίσουμε την δουλειά στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος και φαντάζομαι ότι θα μας έλεγε συνεχίστε να προσπαθείτε να βρείτε καλές λύσεις και να ολοκληρώσετε την επεξεργασία των φακέλων πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ. Και νομίζω μάλιστα ότι αν και ορισμένοι ή ορισμένες από εμά μισούν τη λέξη flexible, οι ίδιοι οι οδηγοί μας ζητούν ένα εύκαμπτο σύστημα για την εργασία και για την ανάπαυση. Και κατά κάποιο τρόπο προκύπτουν και καταστάσεις, όχι μόνο διαφορετικών συνθήκων και διαφορετικών καταστάσεων στις χώρες μέλη, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, όπου ίσως υπάρχει κάποιο ε, ε, πρόβλημα στο λιμάνι ή ε, λόγω του τόπου όπου ε, μεταφέρει κάποια πράγματα ο οδηγός. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζονται πολλές ώρες ευκαμψίας, θα το πω έτσι, 24 ώρες. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να επιτρέπει λίγες ώρες να εργαστεί κανείς με ευφυή τρόπο. Το ίδιο ζητούμενο είναι να είναι λιγότερο γραφειοκρατικό το σύστημα και μικρότερο το βάρος για τον οδηγό με τη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων κλπ. Και κάτι που αποτελεί πρόκληση για όλες και όλους μας σε όλα τα σχετικά ε, θέματα, ε, ανάπαυση, εργασία, καμποτάζ κλπ. Είναι να έχουμε αυτή την κοινή πλατφόρμα δεδομένων με την οποία να συμφωνήσουν όλες οι χώρες μέλη, να μπορεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το πιο σημαντικό εν τέλει σχετικά με την εβδομαδία ανάπαυση είναι κανένας να μην κάνει την εβδομαδία ανάπαυση μέσα στο φορτηγό ο ορισμός της εστίας, του σπιτιού, του home, ποιος θα πει σε κάποιον οδηγό να εδώ αυτό είναι το σπίτι σου όπου μπορείς να αναπάβεσαι. Και αυτό λοιπόν είναι δύσκολη υπόθεση. Το ίδιο πόσο θα πρέπει να πληρώνεται ή τι θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ώστε να μπορέσει ο οδηγός να επιστρέψει σπίτι του. Και τι γίνεται άμα ε, ε, το σπίτι του είναι στις Μπαχάμες ότι ο επιχειρηματία θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση αν υπάρχει η κοινή βούληση. Έμαθα σήμερα ότι ο ευφυής e ταχογράφος για ορισμένους είναι βρισιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπα πρέπει να αποφευθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση και σε βάρος των εταιριών και σε βάρος των επιθεωρητών και των οδηγών. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εργασία αυτή ώστε τα φορτηγά στο μέλλον είναι εξοπλισμένα με τους ευφυείς ταχογράφους που δίνουν πολλές πληροφορίες. και στις περιπτώσεις εκείνες όπου επιβάλλονται ποινές, πρόστιμα, για να βρεθούν αυτοί που έχουν κακή συμπεριφορά και να τιμωρηθούν αυτοί. Αλλά συνήθω, όπως τα πάμε έτσι, θα επιβάλλουμε ποινέ σε όλους, συλλογικά δηλαδή. Σε όλους του φακέλου που έχουμε. Και αυτό με ανησυχεί κάπω, διότι αυτοί που ε, υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις τέλος πάντων και πλαστογραφούν τα δεδομένα, τους έχουμε μπροστά μας την πραγματικότητα και δεν καταφέρνουμε ωστόσο να τους βρούμε και να τους ε, κατονομάσουμε. Ελπίζω ότι θα έχουμε χρόνο λοιπόν για να εκπονήσουμε τέτοιες λύσεις που θα επιτρέπουν να επιβάλλονται ποινές, πρόστιμα σε αυτούς που το αξίζουν και όχι σε όλους, όπως συνήθως κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Κίλονεν. Ο κύριος Ζιλούχ. Ζήλε. Δεν προλαβαίνω δύο επιτροπές ταυτόχρονα κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη που καθυστέρησα. Πρώτον, ευχαριστώ ΒΙΜ για την δουλειά που κάνεις. Είμαστε επιφυλακτικοί και αυτή είναι η ομάδα, αυτή είναι συγγνώμη, η άποψη της ομάδας μας. Είμαστε κατά της ρύθμισης για τα ελαφρά οχήματα. Για την επιστροφή στο σπίτι να το κάνουμε πιο εύκολο αυτό, όπως είπε και ο εισηγητής στην αρχή, γιατί ό,τι και να προσπαθήσουμε να βρούμε, δηλαδή αν είναι ο τόπος της έδρας, ο τόπος της καταχώρησης και ταξινόμησης του αυτοκινήτου, είναι δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του όπου επιθυμεί. Και γι' αυτό ας παραμείνει στην προσωπική επιλογή του οδηγού. Οι περισσότεροι ωστόσο δεν ενδιαφέρονται οι εργοδότες δηλαδή, δεν ενδιαφέρονται οι περισσότεροι αν ο εργαζόμενος επιστρέφει σπίτι του. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην εργάζονται στην αγορά της έδρας τους. Γι' αυτό να πρέπει να μείνει στη συμφωνία μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη. Αυτό είναι εντάξει. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε, εν πάση περιπτώσει, τα πάντα. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε από το επίπεδο της ευρωπαϊκής Νομοθεσία στη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, στην περίπτωση αυτή δηλαδή του επιχειρηματία και του οδηγού. Ας κάνουμε λοιπόν τη ρύθμιση απλή και ελεύθερη επιλογή του οδηγού, ώστε να μπορεί να περνά τον ελεύθερο χρόνο του όπως επιθυμεί σε συμφωνία με τον εργοδότη του. Τώρα, για το αν θα αναπαύεται μέσα στον ε, θάλαμο του οδηγού, η προσέγγιση του βήμη είναι εντάξει. Θα πρέπει να επιτρέπεται αυτό και ιδίω αν δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι στάθμευσης, το οποίο ήδη συμβαίνει. Η συσσόρευση τώρα του χρόνου εργασίας, εμείς έχουμε πει 4 εβδομάδες και 180 ώρες, δεν μας υποστηρίζει αυτό ο εισηγητής, επανερχόμαστε όμως εμείς για να εκφράσουμε τη θέση μας και θα πούμε γιατί, διότι βεβαίως η Ευρώπη έχει και περιφερειακές χώρες, δεν έχει μονάχα κεντρικές χώρες, ειδικά για, το, για τις μεταφορές ε, οδικά και για την ε, εισαγωγή των εφιών ταχογράφων. Εμείς δεν συμφωνούμε το 2020. Μάλλον κάπου 2026 μας φαίνεται μας πιο σωστό. Ίσως έχουμε κάποια διαφορά με απόψε και μεταξύ μας στην ομάδα των Ευρωπαίων Μεταρρυθμιστών και Συντηρητικών. Ας παραμείνει όμως μέσα στα πλαίσια της ε, διαπραγμάτευσης και στη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Αλλά το 2020 όμως είναι υπερβολικά ε, κοντά, υπερβολικά σύντομο το χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ κύριε Ζήλε. Κύριε Κόχ. Δεν κατάλαβα από τη μετάφραση ότι είχατε πει το δικό μου όνομα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ λοιπόν, Βιμ, για την θαυμάσια έκθεση που θέτει τον δάχτυλο επί των τύπων των Ήλων, όπως συμφωνώ και εγώ. Και πρώτα-πρώτα έλεγχος για την τήρηση των ρυθμίσεων. Τρία ζητήματα έχω εγώ να υποβάλω στην προσοχή σου. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να επεκταθεί και στα ελαφρά φορτηγά οχήματα. Και αυτά που είναι πάνω από 2,8 τόνους μεικτού βάρους. Μικτού βάρους. Διότι πρόκειται για πραγματικούς επαγγελματίες οδηγούς. Αυτοί δηλαδή που οδηγούν αυτά τα οχήματα και που είναι κάτω από τους 3,5 τόνους μεικτού βάρους δεν έχουν αυτή τη στιγμή καμιά ρύθμιση για την εργασία και την, και την ανάπαυση. Προτιμούν λοιπόν πολλοί εργοδότε να τους βάζουν να οδηγούν 2,8 τόνους και όχι 3,5 τόνους. Τώρα, χρόνια ανάπαυσης πρέπει να τηρηθούν απαραίτητο. Δεύτερο, η ρύθμιση των 12 ημερών για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Γιατί πρέπει να περιοριστεί αυτό μονάχα σε διαμεθοριακές και να μην εφαρμόζεται και σε εθνικές μεταφορές. Θα χαρώ πολύ αν στη διάρκεια της διαδικασίας μπορέσουμε να προβλέψουμε εδώ μια διόρθωση. Τρίτο, ευφυείς ταχογράφοι. Να θεσπιστούν πολύ, πολύ συντομότερα από αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ έχω βάλει 2020 στην πρότασή μου. Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει ο ευφυής ταχογράφος να αποτελέσει και νομική προϋπόθεση και για την αδειοδότηση του επιχειρηματία. Διότι όλα αυτά τα πράγματα συνδέονται απολύτως μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η κυρία Λουκασέσκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Βιμ και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Είμαι πεπισμένη ότι όλες οι προτάσεις στα πλαίσια της κινητικότητα είναι δύσκολες και θα χρειαστούν συμβιβασμούς, πολύ αμοιβαία κατανόηση. Έχω εδώ κάποιες παρατηρήσεις να κάνω, γιατί και εγώ έχω καταθέσει τροπολογίες, και να αναφερθώ στα, στους πιστοποιημένους χώρους στάθμευσης. Είπε ο εισηγητής ότι θα μπορεί ένας οδηγός να κοιμηθεί στην καμπίνα. Τι γίνεται, αν δεν υπάρξουν πιστοποιημένοι χώροι στάθμευσης σε όλες τις χώρες, τότε κάνοντα και θεσπίζοντα αυτή την πρόταση, εμείς δημιουργούμε κάποιο χάο, κάποια αταξία σε αυτό το θέμα. Γιατί ούτως ή άλλως αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη και θα πρέπει οι επιχειρηματίες να αναλάβουν το κόστος της ε, διανυκτέρευσης. Τώρα για το θέμα της ανάπαυσης. Δεν θα έπρεπε να έχουμε θέσεις άτεκτες για αυτό το θέμα. Όλοι μας γυρνάμε στο σπίτι μας και ο ίδιος ο οδηγός θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να αναπαυθεί στο σπίτι του ή όχι. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία στα πλαίσια της εβδομαδιαίας ανάπαυσης μέσω ας πούμε της συντόμευσης ή της ισόρευσης αυτού του χρόνου στις εβδομάδες και πώς θα το υπολογίζουμε αυτό. Νομίζω ότι ίσως αυτή την περίπτωση αν έχει η οικογένεια, είναι η οικογένεια έχει πραγματικά οδηγό, θα μπορούσε να πάει στην οικογένειά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρώτο και τελικό λόγο εσά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα, Θεωρώ ότι το σχέδιο είναι σωστό, είναι ισορροπημένο, έχει τη σωστή εστίαση και συμφωνώ. Μόνο δύο-τρία επιμέρους σημεία να τονίσω για τροφή για σκέψη περισσότερο. για τους ευφυείς ταχογράφους. Ποιο το σκεπτικό εδώ και ποια είναι η προστιθέμενη αξία σε σχέση με τους τωρινούς ταχογράφους, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές επιπτώσεις της θέσπισης αυτών των ευφυών ταχογράφων. Κοιτάξαμε και ελέξαμε πραγματικά αν μπορούμε να εξοπλίσουμε όλα τα φορτηγά με εφηείς ταχογράφους μέχρι το 2020. Κύριε Κράμερ, ένα λεπτάκι, δεν τέλειωσα ακόμα, περιμένετε λίγο. Γιατί μήπως θα έπρεπε να πούμε ότι εντάξει, να κάτσουμε να δούμε σε περίπτωση προβλήματος σε τι μας εξυπηρετεί ένας εφηείς ταχογράφος. Αν το κάνουμε αυτό, πρώτα, ίσως να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αλλιώς δεν ξέρω. Νομίζω ότι η τωρινή ταγογράφη είναι μια χαρά. Τώρα και σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε ας έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Δεύτερο σημείο για την ανάπαυση και το χρόνο ανάπαυσης στην καμπίνα. Να δούμε τι γίνεται με τις υποδομές. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει μια δικασία παραβίασης της Κομισιόν που σήμερα σε σχέση με χώρες οι οποίες έχουν την υποχρέωση για ανάπαση κάθε 150 χιλιόμετρα. Για, για ποιο λόγο δεν συμβαίνει αυτό. Το να έχουμε μια απαγόρευση χωρίς παρεκκλήσεις, αυτό είναι ο ευκολότερος τρόπος να προστατεύσω την αγορά μου. Οπότε αυτές οι τροπολογίες που προβλέπουν ακριβώς εξαιρέσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πάντως, γενικά θεωρώ θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να λειτουργεί σωστά, έστω και αν έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, θα πρέπει όλοι να στοχεύουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί σωστά στην αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αγιαλά Σεντέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. να ευχαριστήσω τον κύριο Βαντεκάμπ για τις δυνατότητες που μας δίνει. Εμάς στις χώρες της περιφέρειας μας ενδιαφέρει στον υπολογισμό των τεσσάρων εβδομάδων να υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας για τον υπολογισμό της εβδομαίας ανάπαυσης για να μπορούν να πάνε σπίτια τους οι οδηγοί γιατί αυτό θέλουν. Αντί να μένουν σε κάποια πάρκινγκ ανασφαλή, χωρίς ασφάλεια στη Γαλλία ας πούμε. Μετά για τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης, μακάρι να είχαμε αρκετούς πόρους και τη δυνατότητα να πείσουμε τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες ώστε να υλοποιηθούν αυτή η ασφαλείς χώρη στάθμευσης. Πάντως, από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα για τους οδηγούς, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Να μην χρειάζεται δηλαδή να γίνει διάρθρωση στο τομέα και απολύσεις και ανεργία. Επίσης για τον ευφυή ταχογράφο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέπετε η δυνατότητα καταγραφής διέλευση των συνόρων, αυτόματης διέλευση των συνόρων, ώστε να μην τιμωρείτε ή να μην ζημιώνεται ο οδηγός κάθε φορά περνάει τα σύνορα. Μετά για τις κυρώσεις, θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη μας την ανάγκη να υπάρχει κάτι τέτοιο, όμως στο πλαίσιο της Ένωσης. Δηλαδή, θα θέλαμε να μην υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα, η διμερής που υπήρξε σε κάποιες περιπτώσεις. Να υπάρχει κάτι δηλαδή το οποίο θα είναι ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές. Και νομίζω θα ήταν καλό να στοχεύσουμε τελικά μια μέρα σε μια ευρωπαϊκή αρχή η οποία θα μπορούσε να αξιολογήσει και να υποπτεύσει όλο τον μηχανισμό και την εφαρμογή του. Διαφορετικά θα επανέλθουμε σε καταστάσεις όπου θα ανακύψουν ερμηνείες και εφαρμογές διαφοροποιημένες μεταξύ δηλαδή χωρών ε, διέλευσης και χωρών της περιφέρειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαντέρ. Κύριος Δρικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για αυτή την ισορροπημένη έκθεση για ένα λεπτό ζήτημα. Δύο σχόλια, ένα γενικό και ένα ειδικό. Γενικά πρώτα. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς ότι θα πρέπει να αποδεχτεί μια υποβάθμιση των συνθήκων εργασία του. Οπότε όταν μιλάμε για ευελιξία να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί η κοινή γνώμη προσδοκά εμείς να βελτιώσουμε συνθήκες, όχι να τις υποβαθμίσουμε. Και μετά επιμέρους παρατήρηση για τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης γιατί γύρω από αυτούς τους χώρους ε, στάθμευσης συζητάμε και θέματα όπως η ανάπαυση, η χρόνος ανάπαυσης, ανάπαυση στην καπίνα κτλ. Αναφέρεται πολύ αυτό το ζήτημα λοιπόν. Το πρόβλημα δεν είναι να τα φτιάξουμε αυτά τα πάρκινγκ, τα ασφαλή, αλλά να τα λειτουργήσουμε, γιατί κοστίζουν πολύ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει προσωπικό φύλαξης. Βίντεο επιτήρηση κλπ. Οπότε η λειτουργία τους απλά και μόνο σημαίνει ότι δεν είναι δωρεάν η πρόσβαση, πρέπει κάποιος να πληρώσει. Να πληρώσουμε λοιπόν τη στιγμή που δεν μπορούμε καν να τους φτιάξουμε αυτούς τους χώρους, αδύνατο. Και μάλιστα υπάρχουν ελάχιστοι χώροι ασφαλής, χώροι ασφαλής χωρίς γιατί κανείς δεν θα πλήρωνε. Οπότε, αν καταφέρουμε να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα, δηλαδή να φτιάξουμε αυτού του χώρου και να καθορίσουμε τα κόστη λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πληρωμή. Γιατί δεν θα πληρώσει ο ίδιο ο οδηγό την πρόσβαση και χρήση αυτών των ασφαλών χωρών στάθμευση. Οπότε θα πρέπει ο εργοδότη ο... να πληρώσει δίνοντας στον οδηγό κάποιο ποσό σε σχέση με τις προβλεπόμενες τάσεις και σταθμεύσεις. Αλλά μέχρι τότε θα, θα συνεχίσουν οι οδηγοί να, ή θα μπορούσαν οι οδηγοί να παρκάρουν σε χώρους μη ασφαλής για να κρατήσουν τα χρήματα αυτά. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος λειτουργίας αυτών των ασφαλών χωρών στάθμευσης αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παληθεύουμε την χρήση και παραμονή σε αυτούς τους χώρους εκ μέρους των οδηγών ώστε να δουλεύουν σωστά. Από τη στιγμή λοιπόν που θα έχουμε ένα τέτοιο σωστό σύστημα λειτουργία, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με τη λειτουργία και δημιουργία καταρχάς αυτών των ασφαλών χωρών στάθμευση. Αν δεν υπάρξουν αυτοί οι χώροι τότε θα βρεθούν άλλες ε, λύσεις ε, πιο ακραίες. Υπάρχουν θερμάσεις βέβαια καμπίνες ε, στα φορτηγά. Αλλά οι περισσότερες καμπίνες δεν ενδείκνυνται. Έστω και να υπάρχουν κάποιες και μεντούς κιόλας. Τελικά υπάρχει ο κίνδυνος λοιπόν να μην υπάρχουν ασφαλείς χώροι στάθμευσης και οι λίγοι που θα υπάρχουν δεν θα λειτουργούν σωστά. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Ρομπονταλόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο φάκελος και πρέπει να το χειριστούμε με μεγάλη σοβαρότητα. Σε ό,τι φορά την ε, ανάπαυση στην καμπίνα θα ήθελα να, να πάρουμε λίγη απόσταση και να εξετάσουμε το εξή ερώτημα. Πραγματικά τον 21ο αιώνα είναι τόσο δύσκολο για μια εταιρεία μεταφορών να οργανώσει ε, την ανάπαυση των ε, εργαζομένων τη ώστε μέσα σε 14 ημέρες να λάβουν οι οδηγοί ανάπαυση 45 ε, ώρων εκτός καμπίνας. Από τις 24 ώρες στην καμπίνα θέλουν να πέσουμε, το οποίο δημιουργεί ευελιξία και για την επιχείρηση. δεν γίνεται για εβδομάδες και εβδομάδες να ε, αναγκάζουν οι επιχειρήσεις, τους εργαζομένους να αναπαύονται μέσα στην καμπίνα. Είτε πρόκειται για ε, χώρους στάθμευσης είτε όχι, ε, έτσι και αυτοί οι χώροι στάθμευσης υπάρχουν ήδη, απλώς δεν χρησιμοποιούνται επειδή πρέπει να καταβληθεί αντίτιμο. Θέλουμε την τροποποίηση τη περίοδου αναφορά από τι 2 στι 4 εβδομάδε. Έχουμε καταθέσει τροπολογίε για την μέγιστη, το μέγιστο χρόνο οδήγηση στην εβδομάδα. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και πρώτα, για τον κύριο Κοχ. Προ 15 ετών ήδη είχαμε διαφωνήσει για τους ταχογράφους και κάθε φορά λέμε «Α, ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα». Όχι, έχει έρθει η ώρα. Φτάσαμε στην ψηφιακή εποχή. Και νομοθεσία χωρίς έλεγχο, έχει εκεί δίκιο ο Βιμ δεν γίνεται τίποτα. Το απλούστερο και το φθηνότερο είναι να γίνει η δουλειά αυτή με τους ταχογράφους. Και ο εξοπλισμός των φορτηγών μέχρι το 2020 δεν είναι και πολύ. Αν συμφωνήσει ο κλάδος και γνωρίζουν μέχρι το 2020, θα δείτε πόσο θα επιταχυνθεί η διαδικασία. Είχαμε και την υπόθεση με τον εξοπλισμό κατά του θορύβου. Όταν έφτασε η ώρα, ξαφνικά εμφανίστηκαν 6-7 επιχειρήσεις και τώρα 80% των ε, εμπορευματικών βαγονιών στο σιδηρόδρομο είναι εξοπλισμένα με τους μηχανισμούς αυτούς. Μετά είπε κάποιος άλλος συνάδελφος ο οδηγός να αποφασίσει εάν θα πάει σπίτι του να ξεκουραστεί ή όχι. Ωραίο θα ήταν, αλλά δεν αποφασίζει ο οδηγός. Όταν είχαμε πάει στους σταθμούς ελέγχου, μας είπε ένας αστυνομικός, ναι, χθες λάβαμε ένα τηλεφώνημα και κάθε μέρα μάλιστα ένας οδηγός φορτηγού μας είπε σας παρακαλώ ελάτε να με ελέγξετε είμαι ήδη 17 ώρες στο τιμόνι χωρίς, ε, χωρίς διάλειμμα δεν μου επιτρέπει το αφεντικό να τηρήσω τους ε, χρόνους ανάπαυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι πολύ επικίνδυνες και όχι μόνο για τον οδηγό αλλά για όλους που κυκλοφορούν στον δρόμο. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά τα πράγματα αυτά. Ο μόνος τρόπος είναι να γίνει αυστηρή επιβολή του χρόνου αναπαύσεως και μάλιστα αυτό γίνεται μόνο με τον ταχογράφο. Σε ό,τι αφορά τους τελέχους, σήμερα το βράδυ υπάρχει εκδήλωση του Βιμ και άκουσα εγώ ότι υπάρχουν, έγινε ένας καυγάς, διότι μάλωσαν μεταξύ τους για τον χώρο στάθμευσης. Γίνονται ελεγχοί. Στο Βέλγιο και στις κάτω χώρες γίνονται 80% έλεγχοι. Και είναι αυστηρά τα πρόστιμα. 500 ευρώ για τον οδηγό, 1500 για την επιχείρηση. Σύγκριση τώρα με τη Γερμανία. Είναι καταστροφή. Ακόμα και όταν γίνονται έλεγχοι δεν γίνεται τίποτα. Τους κάνουν μια μικρή επίπληξη και τελείωσε. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή ισχύω κανόνα. Δεν επιτρέπεται να γίνουν τα πράγματα αυτά, ενώ πάντα την ανάπαυση των οδηγών. Αυτό είναι όχι μόνο για το συμφέρον του οδηγού, αλλά και για το συμφέρον της τροχέας ασφάλειας. Πρέπει να φανούμε πολύ αυστηρότεροι και τα δικαιώματα αυτά πρέπει να ισχύσουν πανευρωπαϊκά. Ευχαριστώ. Κύριε Κράμερ, δεν έχω άλλον κανένα γραμμένο, λέει η πρόεδρος Ντελή. Τώρα, η κυρία Βέρνερ της Κομισιόν. Μιλούμε και για ομολογάρισμα των ε, εξοπλισμών για την διάβαση των συνόρων. Τι θα μας πείτε γι' αυτό. Να μας απαντήσετε κυρία Βέρνερ για όλα τα θέματα, χώρους σταθμεύσεως και ούτε καθεξής. Πού βρισκόμαστε και σχετικά με την απαγόρευση αναπαύσεως ε, μέσα στο θάλαμο του αυτοκινήτου. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ αυτή ζωντανή συζήτηση και την ιδιαίτερα εξορροπημένη πρόταση στην έκθεση του κυρίου Βαντερκάμπ. Υπενθυμίζω ότι σκοπός ε, της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στην αρχική προσέγγιση ήταν ε, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ανταγωνισμού και των εργασιακών συνθήκων με εξισορροπημένο τρόπο, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι έχουμε και δυνατότητες ενισχυμένης και ευφυού επιβολής του νόμου, που είναι αυτό που μας λείπει σήμερα. Προφανώ και υπάρχουν πολλέ τροπολογίε για αυτή την πρόταση. Είναι ε, σημαντικό το ενδιαφέρον και ο κύριος Βαντερκάμπ έχει εντοπίσει τις βασικές ενότητες. Πρώτον, έχουμε την έννοια της απαγόρευσης ε, της ανάπαυσης στην καμπίνα. Αυτό ήταν ένα τμήμα της ε, πρότασης της Κομισιόν. Και η, απόφαση, η συζήτηση είναι σημαντική. Λέμε δηλαδή ότι υπάρχει γενική απαγόρευση εκτός και αν το φορτηγό έχει σταθμεύσει σε ασφαλή χώρο στάθμευσης. Και μετά περνάμε στη συζήτηση τι συνιστά ε, ασφαλή χώρο στάθμευσης, ποιος το ορίζει, ποιος το πιστοποιεί. Νομίζω ότι με καλή θέληση ε, μπορούμε να καταλήξουμε σε μία ε, σωστή λύση και λίγο πιο περίπλοκο ζήτημα πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα ε, δημιουργούνται, θα κατασκευάζονται και θα λειτουργούν αυτοί οι χώροι στάθμευσης σε επαρκή αριθμό και πυκνότητα σε όλη την Ευρώπη. Και μετά υπάρχει και μία ε, συζήτηση γλωσσολογικού ενδιαφέροντος, ε, μήπως ε, τα διόδια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους σταθμούς και κατά πόσο υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών, η οποία προκύπτει από την νομοθεσία για τα δίκτυα TNT ή κατά πόσο θα πρέπει να λειτουργούν με, σε εμπορική βάση αυτοί οι σταθμοί. Γιατί εάν είναι να επιβάλλουμε απαγόρευση, τότε θα δημιουργήσουμε και ζήτηση ε, για τους ε, οδηγούς. Να χρησιμοποιούν δηλαδή αυτού του σταθμού. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να παράσουμε όλε τι τεχνικέ λεπτομέρειε που έχουμε στη θέση σα και νομίζω ότι ήδη σα ενημέρωσα ότι χάρη σε ορισμένα πιλωτικά έργα που πρότεινε ο κύριος Βαντάλε, εκπονείται τώρα μία ε, μελέτη για αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς τα αποτελέσματα θα τα έχουμε μόνο στη συνέχεια της χρονιάς. Τώρα, η επιστροφή στην αιστεία. Και από τη σημερινή συζήτηση προκύπτει ότι παρότι αυτό είναι κάτι το θετικό για τις εργασιακές συνθήκες του οδηγού, είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς ε, το τι είναι αιστεία, το σπίτι δηλαδή. Είναι λίγο υποκειμενικό, εξαρτάται από τον ορισμό. Από τη δική μας πλευρά, ο εργοδότης θα πρέπει να οργανώνει έτσι το πρόγραμμα του οδηγού, ώστε να είναι σε θέση να επιστρέψουν ενδεχομένως στην ε, έδρα ή στο, κέντρο επιχειρήσεων του εργοδότη ή στην, στο χώρο διαμονής, ε, στην κατοικία δηλαδή, να επιστρέψει στην κατοικία του ο οδηγός. Είναι μία από τις δύο λύσεις. Συμφωνούμε επίσης με τον εισηγητή ότι θα πρέπει κάποια ευελιξία να δώσουμε ε, για την επιστροφή στην αιστεία ως προς τον χρόνο οδήγησης. θα πρέπει δηλαδή να υποχρεώσουμε τον οδηγό να ε, πάρει την εβδομαδιαία του ανάπαυση σε ένα χώρο στάθμευση που είναι πολύ κοντά, μερικά χιλιόμετρα το σπίτι του, επειδή ε, δεν μπορεί να υπερβεί τον συνολικό χρόνο οδήγηση. Μετά, για τον ευφυή e ταχογράφο και τις ημερομηνίε. Να ξεκαθαρίσω ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μεγάλο ενθουσιασμό ε, αυτή την πρόταση, δηλαδή να ισχύει σε αυτό το μέτρο πιο νωρίς. Δεν κάναμε πρόταση από αυτού. Πρόκειται για, τον, για την ισχύουσα νομοθεσία που έθεσαν ε, τόσο μακριά στο μέλλον αυτή την ημερομηνία. Εμεί με τα χαρά να τη φέρουμε πιο κοντά. Και υπήρξε όντω και μια συζήτηση στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου για ορισμένα ε, σχετικά ζητήματα. Τρία θέματα εξετάσαμε στο Συμβούλιο. Πρώτον, η επέκταση της περίοδου για τους ε, ελέγχου στο οδικό δίκτυο και τα δεδομένα που θα πρέπει να καταγράφονται στον τοχογράφο. Μετά η καταχώρηση της διάσχησης των συνόρων και αυτό τι σημαίνει για τη δυνατότητα της κάρτας και τη χωρητικότητα μάλλον της κάρτας ε, και κατά πόσο μπορεί να ε, καταγράψει τη διέλευση των συνόρων και για την αναδρομική ισχύ, το retrofit, έχουμε λάβει την πρώτη εκδοχή της μελέτης ε, για αυτό το ζήτημα, η οποία μας δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα. Φυσικά και θα σας ενημερώσουμε απευθείας μόλις ε, δημοσιευθεί, όμως ε, τα προκατακτικά πορίσματα, και αυτό είπαμε και στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, μας δείχνει λοιπόν η μελέτη μία εικόνα των οχημάτων που θα πρέπει να τύχουν αυτής της προσαρμογής και τα εργαστήρια που απαιτούνται και το κόστος. Το κόστος του τοχογράφου είναι περίπου 1000 ευρώ, αλλά έχουμε χρειαζόμαστε ακόμα περίπου 1.000 ευρώ για την εγκατάσταση, την κατάρτιση του οδηγού για το εργαστήριο αυτό και η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι συνολικά περίπου 2026 το 2026 είναι μια ρεαλιστική ημερομηνία για την θέση σε σχέση του μέτρου. Φυσικά και ε, αυτά τα εργαστήρια δεν είναι είναι προκαθορισμένα, αλλά δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής βούλησης, υπάρχουν και αντικειμενικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Να πω και κάτι για την επιβολή του νόμου και την πρόσβαση ε, στη πληροφορία. Ανταλλαγή πληροφοριών, είπατε, μεταξύ εθνικών αρχών. Αυτό πραγματικά είναι κέρια σημασία για να υπάρξει και σωστή επιβολή του νόμου. Και εμεί θεωρούμε ότι το σύστημα ενίας αγοράς που ήδη υπάρχει ε, είναι ένα πολύ καλό μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διοικήσεων και για να αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις. Όταν υπάρχει ήδη ένα ισχύον σύστημα, δεν χρειάζεται να βρούμε δεύτερο. Τώρα, ξέρετε, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Μαρτίου υιοθέτησε μια νέα πρόταση για μία αρχή που θα μπορούσε να είναι ιδίως ιδιαίτερως δραστήρια και στις οδικές μεταφορές. Θέλουμε να ε, εργαστούμε περαιτέρω σε αυτή τη δομή και προσβλέπουμε και στη στήριξη του Κοινοβουλίου. Δύο ενότητες ε, τροπολογιών ε, προσθέτουν νέα στοιχεία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να τις εξετάσουμε με θετικό μάτι και είμαστε, είμαστε να βρούμε μια καλή λύση. Η ευελιξία για τους οδηγούς λεωφορείων και πούλμαν που όντως ε, βρίσκονται στη διαφορετική κατάσταση από τους οδηγούς φορτηγών και για να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε υπόψη στην ομοθεσία τα αυτόνομα οχήματα. Σε ό,τι αφορά και τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Τέλος, τα ελαφρά εμπορικά οχήματα. Η Επιτροπή είναι υπέρ της επαγγελματοποίησης του κλάδου, αλλά είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε και μια αναλογική προσέγγιση. Η εφαρμογή των κανόνων για την πρόσβαση στο επάγγελμα είναι ένα πρώτο αλλά δεν είναι σκόπιμο αυτή τη στιγμή ε, να υπάρχει προϋπόθεση εγκατάστασης ταχογράφου σε αυτά τα οχήματα. Και πράγματι Υπάρχει μια ευελιξία για το ακριβές βάρος των οχημάτων που θα καλύπτονται από τις διατάξεις, αλλά θα επανέλθουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Merci, Madame Werner. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαντερκάμπ. Συμπερασματικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι πολλοί μας ακούν και μας βλέπουν σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σταθώ έτσι ε, περαιτέρω σε ορισμένα στοιχεία. Το πρώτο που ανέφερε η κυρία Μάισνερ, η οποία δυστυχώ έπρεπε να αποχωρήσει. Η χρήση του ταχογράφου στα ελαφρά εμπορικά οχήματα. Σε ό,τι αφορά το κράτος μέλος, εθνική χρήση δηλαδή. Εάν κάποιος οδηγεί από το Μόναχο στο Αμβούργο, είναι, δεν καθόλου περίεργο να ελέγξει κανείς ε, ε, τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, γιατί πρόκειται για τεράστια απόσταση. Το ίδιο και αν κάποιος πηγαίνει από το Παλέρμο στο Μιλάνο. Και πάλι είναι καθόλου λογικό να ελέγξει κανείς τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Και αυτό ε, αναφέρθηκε και στη τελευταία συνεδρίαση των σκιωδών, ότι δημιουργεί όντως ε, σημαντικό θέμα εδώ. Και με ενδιαφέρει ιδιαίτερος αυτό, να το πω απευθεία ε, στα συνδικάτα. Για αυτά που είπε ο κύριος Τέιλορ. Σίγουρα και υπάρχει μεγάλη συνάφεια μεταξύ αυτού του φακέλου με το φάκελο της απόσπασης και του καποτάζ. Και χαίρομαι που είναι εδώ ο Ισμαήλ θέλουμε να τα συσχετίσουμε αυτά τα τρία συζητήματα. Γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Πρέπει να υπάρχει μια καλή συνέργεια μεταξύ των τριών αυτών φακέλων. Μετά, Πρόεδρε, ο Παβέλ Τελίτσκα έκανε δύο σημαντικές παρατηρήσεις που κάπως πλαισιώνουν και τη συζήτηση. Εγώ προσωπικά μένω στο Less regulation, better digitalization. Λιγότερη νομοθεσία, περισσότερη ψηφιοποίηση. Οι δυνατότητε που μας δίνει η ευφυής e ταχογράφου είναι τεράστιε. Ε, οι εξελίξει είναι ραγδαίες. Βλέπετε τι γίνεται με την ψηφιοποίηση στην Κίνα, στην Ινδία, στι ΗΠΑ. Δεν γίνεται εμεί να μείνουμε πίσω. Και βέβαια, αυτή η ευφυή e ταχογράφη σύντομα θα, λάβουν, ε, θα εξοπλιστούν και με GPS. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Θα ξέρει λοιπόν ακριβώ πού είναι το φορτηγό και πότε ε, περνάει τα σύνορα. Θα έχουμε και αυτό το ίδιο στοιχείο. Όλα αυτά τα δεδομένα καταγράφονται από τον τοχογράφο. Και εδώ, Πρόεδρε, είναι σημαντικό να έχουμε σαφή νομοθεσία. Γιατί τότε θα ακολουθήσει και η αγορά. Αν εμεί πούμε καλά, εντάξει, δεν πειράζει, κάντε ό,τι θέλετε. Ε, και το 2029 ξαναβλέπουμε τότε δεν θα μας ακολουθήσει η αγορά. Οπότε, σε αυτό επιμένω πραγματικά. Άκουσα με προσοχή τα άσοπη κυρία Βέρνερ για το retrofitting, τη μετατροπή των φορτηγών. Όμως αυτό το κόστος δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο και δικαιολογία για να αναβάλουμε πάπυρον την εγκατάσταση των ε, ταχογράφων γιατί είναι απαραίτητο εργαλείο για τον ε, για τη διασφάλιση του χρόνου ανάπαυσης των οδηγών. Η δεύτερη παρατηρήση του Παβέλ Τελίτσκα για την απαγόρευση της ε, ανάπαυσης στην καμπίνα. Ε, εντάξει, είναι πολύ εύκολο για τη Γαλλία και τη Γερμανία να πούν ότι εμείς δεν θα εφαρμόσουμε την ανάπαυση στην καμπίνα. Αλλά τότε έχουμε πολλά κοινωνικά προβλήματα στις εθνικές οδούς. Βλέπετε σε πολλές χώρες ότι από πολλές χώρες έρχονται στις κάτω χώρες αυτοί οι οδηγοί γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούν να μείνουν στην καμπίνα στη Γερμανία και στην Γαλλία. Και εδώ να πω και στον συνάδελφο ότι εδώ είναι ο συνδυασμό και ο συντονισμό. Αν υπάρχουν επιχειρήσει που λένε ότι εμεί δεχόμαστε ε, την ανάπαυση στην καμπίνα, θα πούμε εμεί εντάξει, αλλά πρέπει να είναι σε προστατευμένο και ασφαλή χώρο στάθμευση. Η γερμανική κυβέρνηση την 1η Ιανουαρίου 2018 υιοθέτησε και εφάρμοσε ένα ε, ε, σύστημα επιδοτήσεων για χρόνο ανάπαυση σε χώρο στάθμευσης και αυτό κοστίζει 4,18 ευρώ στον οδηγό. Τα υπόλοιπα επιδοτούνται από την γερμανική κυβέρνηση γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορούν να καταπολεμήσουν αυτό το κοινωνικό πρόβλημα με μια στήρα απαγόρευση. Βέβαια, προ τον κύριο Ρικέ, να πω ότι όντω πρέπει να υπάρχει εμπορική λειτουργία αυτών των χώρων στάθμευση. Και γίνεται αυτό. Ποιο θα το πληρώνει, ο, ο εργοδότης. Με ποιον τρόπο, με μια προπληρωμένη κάρτα. Δεν θα δίνουμε πλέον μετρητά, γιατί είναι πολλοί οι ε, οδηγοί που βάζουν αυτά τα χρήματα στη τσέπη για να στείλουν την κόρη του στο πανεπιστήμιο και πηγαίνουν σε έναν ε, αφύλακτο χώρο στάθμευση. Όχι, δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς. Αν θέλει κάποιος να αναπαυθεί ε, στην καμπίνα, θα το κάνει σε έναν χώρο στάθμευσης. Τέλος, για τις παρατηρήσεις της Κριστίν. Σωστά όλα αυτά. Ε, Ένας σωστός εργοδότης ε, αφήνει τους οδηγούς να επιστρέψουν μια φορά στις 14 μέρες στην έδρα τους. Αλλά ο Ρόμπερτ Ζήλε τι είπε πριν προηγουμένω ότι εντάξει, αν κάποιο έρχεται από την Εστονία ή από την Νότια Ισπανία, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Και να υπενθυμίσω στην Κριστίν ότι αν κάποιο είναι στον δρόμο 14, δρόμου, 14 ε, μέρες, ε, πρέπει να δούμε τι θα κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο που έχει. Μπορεί κάποιο να πει εντάξει, θα το στείλουμε σε ένα ξενοδοχείο. Αλλά αυτό είναι μια φτηνή σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση. Πρέπει να εξετάσουμε την πραγματικότητα και για τον εργοδότη και για τον οδηγό. Α, ναι. Και κάτι τελευταίο. Για, την, για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας, τον ELA. Για το ΕΛΚ αυτό είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Εγώ είμαι θετικά διακείμενος, προσωπικά. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εν ώψη των εκλογών του 19 για να δείξουμε ακριβώς ποια είναι η στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς ε, τον ELA. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάμπ. Ευρωπαϊκός οργανισμός που θέτει θέματα, ε, που συζητεί θέματα εργασίας δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα εργασίας των οδηγών. Άρα αυτός ο οργανισμός θα πρέπει να εξετάσει τι γίνεται αύριο και στις οδικές μεταφορές. Οδικέ μεταφορές βέβαια, συνεχίζει η και θα μιλήσουμε και για τι αεροπορικέ μεταφορές με το σχετικό πακέτο μέτρων και βεβαίω και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα τώρα που είναι η έκθεση της κυρίας Κίλονεν για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Ορίστε κυρία Κίλονεν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει να αναζητήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία και στην ελεύθερη διακίνηση ή κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων, δηλαδή στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, όπου πρέπει να υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών και για να γίνουν αυτά χρειαζόμαστε αναλογικούς και καλά αιτιολογημένους κανόνες που να μην προκαλούν περιττό γραφειοκρατικό άχθος, Ιδίω για μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Πρέπει να αυξήσουμε την ελκυστικότητα του, οδηγού, του επαγγέλματος του οδηγού. Α, αστεία πράγματα δηλαδή, βεβαίως όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ εύκολες ε, αυτές οι απαντήσεις. Ορισμένα θέματα που έχουμε ήδη εντοπίσει και όπου φαίνεται να διαμορφώνεται συνένεση στη βάση των, ε, της εξετάσεως των τροπολογιών, ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων απατών, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών και πιο αποτελεσματική συνεργασία, ακόμη και από αυτήν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάγκη να υπάρξει ενιαία θηρίδα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την βελτίωση του συντονισμού, ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν την εργασία μας στην βάση του ΙΜΗ που είναι το Διεθνές Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών Αγοράς να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο Συμβουλίο Υπουργών ότι οι χωρισμένοι δηλαδή υπάρχει ανάγκη να επιταχύνουν την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής ε, διαβίβασης ε, πληροφοριών με τα διάφορα συστήματα, η ΕΟ και ECMR, ανάγκη να υπάρξουν ξεκάθαροι κανόνες και ενιαία εφαρμογή και αυστηρή επιβολή με πάντα χαμηλή γραφειοκρατία. Ανάγκη να επιταχυνθεί η εισαγωγή των εφιών ταχογράφων να υπάρχουν κοινού μορφότυπου έντυπα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάζεται, μάλλον φαίνεται πως συμφωνούμε ότι η έλεγχη του χρόνου εργασίας θα πρέπει να μην γίνονται στις οδούς αλλά στις έδρες των επιχειρήσεων πριν να υπάρξει κάποιο ε, δίκαιο και ε, ευέλικτο σύστημα, διαρκής αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενημέρωσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων. Οι τροπολογίες που έχουν σχέση με τα θέματα αυτά ε, έχουν διάφορες ε, κατευθύνσεις και στη βάση των τροπολογιών φαίνεται ότι το ερώτημα παραμένει ανοιχτό για το εάν ναι ή όχι οι κανόνες απόσπαση εργαζομένων είναι ο, το καλύτερο μηχανισμό για να λυθούν τα σχετικά προβλήματα στι διεθνεί μεταφορέ. Έχουμε λάβει τροπολογίε οι οποίε προτείνουν εναλλακτικά οριζόντια μέτρα στο Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο για να πάυσουν ορισμένες αυθαίρετες πρακτικές και για τις διάφορες κατηγορίες των τροπολογιών μπορούν να ταυτοποιηθούν ότι είναι σε σχέση με τις διεθνείς μεταφορές. Η πρώτη είναι να αποκλειστεί, να αποκλειστούν οι διεθνείς μεταφορές από το καθεστώς απόσπαση εργαζομένων. Δεύτερο, οι διεθνείς μεταφορές να ρυθμιστούν από την πρώτη μέρα. Τρίτο, να, ξεκαθαριστούν ορισμένα θέματα. Και τέταρτο, να ε, φύγουμε από την πρόταση Επιτροπής για το τρίμέρο. Έχουμε και άλλες προτάσεις από μία σε 16 ημέρες και για το καμποτάζ από μία σε 10 ημέρες. Όλοι φαίνεται να συμφωνούμε ωστόσο στο ότι η διαμετακόμιση δεν είναι κατάσταση όπου ισχύει απόσπαση θα χρειαστεί να δουλέψουμε πολύ μετά τις διακοπές του Πάσχα για να επιτύχουμε λύσεις και για τους οδηγούς αλλά και για τις εταιρείε μεταφορών και για τους άλλους φορείς μέσα στην αλυσίδα της εφοδιαστικής. Σημαντική λοιπόν πρόκληση αυτή για μας και ενθαρρύνω όλους και όλους να αναζητήσουν ευφυείς, αν και ο δεν αρέσει η λήξη αυτή, ευφυείς λύσεις λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε τα μυαλά μας, καινοτόμες λύσεις στο κατάλληλο, ε, να, που να εξασφαλίσουν το κατάλληλο επίπεδο κοινωνικής προστασίας και αυτά να μην ε, επιφέρουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Υπάρχουν και ορισμένα θέματα που χρειάζονται πιο ανοιχτή συζήτηση, μεταφορά επιβατών, ενδεχόμενα, ενδεχόμενα εκεί να υπάρξει εξαίρεση από τους γενικούς κανόνες. Τα έντυπα που θα πρέπει να έχει η έγγραφα που θα πρέπει να έχει μαζί του οδηγό, για παράδειγμα δελτία ε, μισθοδοσία και άλλα σχετικά. Ορισμένα από αυτά υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Για να υπάρξουν όμως ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να υπάρχει και κοινή πλατφόρμα. Και το ζήτημα της γλώσσας των ε, απαιτουμένων ε, πληροφοριών. Ποιες γλώσσες, πόσες γλώσσες Πού βρίσκεται εδώ η δίκαιη μεταχείριση. Το ίδιο για τους ελέγχους. Θα γίνονται στην επιχείρηση ή θα γίνονται στην άκρη του δρόμου. Και πληροφορίες επίσης για την δήλωση απόσπαση του εργαζομένου και πρόσθετες πληροφορίες ζητούμε εμείς σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής και έχουμε και κάποιες προτάσεις σχετικά με τις διατάξεις ευθύνης για ολόκληρη την, τη, την αλυσίδα της εφοδιαστικής και αυτό είναι σημαντικό θέμα και πρέπει επίσης να συζητήσουμε ακόμη και ενδεχόμενε κυρώσεις και ποινές που να επιβαρύνουν αυτούς πραγματικά το αξίζουν και όχι όλους, να μην επιβαρύνουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Κυρία Πρόεδρε, Αυτά είναι τα πρώτα μου μαγικά σχόλια και περιμένω με μεγάλη χαρά να ακούσω τι θα πούν οι συνάδελφοι σας και οι συνάδελφοί μου όσοι επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μου. Ευχαριστώ κύριε Κίλονεν. Κύριε Ντελή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μεγάλος αριθμός τροπολογιών ε, πολλές από αυτές έχουν θετικό χαρακτήρα, προσπαθούν να μειώσουν τα βάρη των επιχειρήσεων. Υπάρχουν όμως και τροπολογίες με τις οποίες εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω, διότι οι συμφωνίες αυτές το μόνο που κάνουν είναι να ενισχύουν τα προστατευτικά μέτρα ή τα μέτρα προστατευτισμού τα οποία ήδη υπάρχουν και δεν καθιστούν δυνατή τη λειτουργία της αγοράς των μεταφορών. Πρόκειται για ένα θέμα στη συζήτηση του οποίου φαίνεται να αντιπαρατίθεται η Ανατολή με τη Δύση. Στη διάρκεια των συναντήσεων είδαμε τι πρόσθετε τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει μέσω της ε, πρότασής της. Αυτές οι επιβαρύνσεις θα έχουν αρνητικές συνέπειες για όλους τους φορείς της αγοράς μεταφορών. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των φορέων και ιδίω για τις μικρές επιχειρήσεις της Ανατολικής Ευρώπης, διότι ο στόχος μας είναι ένας και κοινό, δηλαδή η διευκόλυνση της κινητικότητας και το να φτάνουν τα αγαθά, τα εμπορεύματα στον τελικό καταναλωτή γρήγορα και φθηνά. Θα αναζητήσουμε δυνατότητες συμβασμού για να μην δυσκολέψουμε το μέλλον των επιχειρήσεων. Είναι πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς την έλλειψη οδηγών που σημειώνεται σχεδόν σε κάθε χώρα μέλος. Θα χρειαστεί να προσέξουμε πολύ στην νομοθετική διαδικασία, ώστε να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα έλθουν να καλύψουν το κενό αυτό οδηγεί τρίτων χωρών και όπου επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα καλύψουν μερίδια της αγοράς. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτέ τι τρίτε χώρε. Οι επιχειρήσει θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να προσλάβουν οδηγούς και μάλιστα και ως ανεξάρτητους ε, επιχειρηματίες. Στην περίπτωση όμως των ανεξάρτητων ε, ε, αυτών ε, επιχειρηματιών ή επαγγελματιών δεν θα εφαρμόζεται η οδηγία. Χρειάζονται λοιπόν, χρειάζεται να αναζητηθούν λύσεις. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, έχουμε μεγάλο αριθμό διαβουλεύσεων που πρέπει να διεξαγαγούμε. Ήδη και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και στην περίπτωση των άλλων πολιτικών ομάδων είναι αναγκαίο να γίνουν διαβουλεύσεις με τους ε, σκιώδεις και με τον εισηγητή ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Κιλόνεν για την έκθεσή της που μας δίνει κάποιες ενδείξεις για το που πάμε και για τις μελλοντικέ λύσεις τουλάχιστον για κάποια θέματα όπως οι διεθνείς μεταφορές που αναφέρει. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει, γιατί ένας από τους στόχους αυτές τη νομοθεσία ήταν ακριβώς το να πετύχουμε μια απλούστευση. ώστε όσο θαυμάσια και να είναι η νομοθεσία, να μην είχε την επαφή της με την πραγματικότητα όπως έκανε η προηγούμενη. Η κυρία Κιλόναν λοιπόν θέλει να διατηρήσει την ελεύθερη κυκλοφορία και να αποφύγει το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αλλά υπάρχει και άλλη μια πτυχή, δηλαδή η αποφυγή των διακρίσεων σε σχέση με τους ελέγχους στο δικό δίκτυο. και ένα κομμάτι των τροπολογιών μας αυτό ακριβώς αφορά. Σήμερα στους Κιώδης το συζητήσαμε και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εξάγονται ταυτόχρονα έλεγχοι και στις εγκαταστάσεις αλλά και στο δικό δίκτυο, στους δρόμους. Και αυτή η τελική, για να, αυτή η τελευταία για να αποφευχθούν οι διακρίσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη βοήθεια των εφιών ταχογράφων και επειδή δεν θα γίνει άμεσα αυτό για τους ταχογράφους όπως είπε και, είπε και ο κ. Βαντερκάμπ να εφαρμόζονται τα συστήματα ήμι και έρου πλατφόρμες που ήδη χρησιμοποιούνται, που ήδη λειτουργούν ώστε να έχουμε τη δυνατότητα με ηλεκτρονικές εφαρμογές γρήγορες να διευκολύνουμε τους ελέγχους στο δικό δίκτυο χωρίς να μπλοκάρονται τα φορτηγά και να παραμένουν στους πλαϊνούς δρόμους των δρόμων και να κάνουμε ελέγχου στα φορτηγά. Το είπαμε και για τα πρόστιμα, για τις κλήσεις με την Ουγγρική Προεδρία. Είπαμε ότι για τη βάση δεδομένων με τους παραβάτες υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς γίνεται με τις επιχειρήσεις κατά πόσο έχουν παραγωγική συμπεριφορά ή όχι. Οι έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να δημοσιεύονται ώστε ακριβώς να αποφεύγουμε τις διακρίσεις. Συμφωνώ με αυτό που λέει η Κομισιόν, δηλαδή θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι και θα πρέπει να υπάρχουν και συμπεφωνημένοι έλεγχοι πανευρωπαϊκά σε επιχειρήσεις. Και για να απευθούν οι διακρίσεις θα πρέπει να είναι δημόσια τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Στην μετρική οδηγία αναφέρθηκε το θέμα της εργασιακής αρχής. Εγώ συμφωνώ με αυτό, αλλά φοβάμαι ότι η εργασιακή αρχή δεν θα κάνει συγκεκριμενοποιήσεις στα πλαίσια της οδηγίας. Γιατί υπάρχουν αλλού ελλείψεις. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια αρχή, δεν θα έλεγα μια υπηρεσία, αλλά μια αρχή τέλο πάντων ευρωπαϊκή οδικών μεταφορών, όπου πέραν του θέματο του θέματος ασφάλειας θα ασχολείται με τον έλεγχο και την εποπτεία όλων αυτών των ζητημάτων που θα εφαρμόσει η τωρινή νομοθεσία στις μεταφορές. Τέλος, για τις αποσπάσεις, συμφωνώ με την κυρία Κιλώνεν. Δηλαδή να μην αφορά τις διαμετακομίσεις αυτή η, ή της χώρες διέλευσης αυτή η απόσπαση. χωρίς νομίζω ότι η κυρία Κιλόνεν λέει να μην επικεντρωθούμε μόνο στην εφαρμογή του καμποτάζ. Εδώ γι' αυτό θα μπορούσα να συμφωνήσω αν δεν ισχύσει για τις διεθνείς ε, μεταφορές και για το καμποτάζ πάλι συγκεκριμένα από τις 0 μέχρι τις πάνω από 10 μέρες, νομίζω ότι τουλάχιστον για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έπρεπε τουλάχιστον να πούμε ότι αυτές οι οποίες δεν βασίζουν το λειτουργικό τους μοντέλο στο καμποτές και το κάνουν περιστασιακά για συγκεκριμένους λόγους, τότε εκεί θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια εφαρμογή πενθυμέρου, κάτι το οποίο είχε αρχικά προτείνει η Κομισιόν. Συμφωνούμε τελικά ότι όσο νωρίτερα γίνει η εφαρμογή και η χρήση του εφηβούς ταχογράφου, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει σε διάφορες επιπλοκές, τόσο περισσότερο θα προχωρήσουν τα πράγματα και νομίζω θα βοηθήσουμε κυρία Χιλόνη στον προχωρήσει αυτή η νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σαντέρ ο κύριος ε, Τόσκι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να σας φάω χρόνο, γιατί πολλά σχόλια που ήθελα να κάνω υπόθηκαν. Να προσθέσω και εγώ τα δικά μου συγχαρητήρια μαζί με αυτά των υπολείπων προς την κυρία Κιλόνεν. Όπως ξέρετε υπάρχουν πολλές τροπολογίες και υπάρχουν πολλές απόψεις και για την ανέβρεση συμβασμού τα ενδεχόμενα δεν είναι πολλά. Πάντως εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να βρεθούν συμβασμοί. Πάντως εγώ προτείνω το εξής. να έχουμε ένα δικό όνομα, ένα λέξη specialis, που θα μπορούσε να αποκλεί ή να εξαιρεί τις μεταφορές από τις αποσπάσεις. Μετά, εξαίρεση για το καποτάζ στις διεθνείς μεταφορές, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παροχής αυτών των πληροφοριών σε όλους τους ενεργούς φορείς στην ενιαία αγορά και εδώ τονίζω και υπογραμμίζω τη λέξη ενιαία αγορά. το μοντέλο ελεγχών των οδικών δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τους οδηγούς να έχουν πάντα μαζί τους ένα πακέτο με έγγραφα και θα πρέπει η έλεγχοι αυτοί να είναι δυνατόν να γίνουν στην έδρα των επιχειρήσεων. Οπότε εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες απλουστεύσεις, διεκπεριώσεις, επιταχύνσεις για να αποφύγουμε το διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος. Μετά, ελπίζουμε όλα αυτά να εφαρμοστούν σύμφωνα με την κοινή λογική. Δηλαδή, μια γεμάτη μέρα εργασίας δεν μπορεί να είναι για έξι ώρε οδήγηση. Τα εξηγούμε όλα αυτά πάντω στι τροπολογίε μα και σα ευχαριστώ πολύ που δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζοντοσκή. Ο κύριο Ντένι Καβό Εκπροσωπείτε την κυρία Μπιλμπάου, ναι. Η κυρία Μπιλμπάου απουσιάζει. Έχει άλλε επίγουσε υποχρεώσει και μου ζήτησε να μεταβάσω κάποιε απόψει της. ευχαριστεί τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε μέχρι τώρα και βέβαια κατανοεί ότι ο φάκελος είναι περίπλοκος. Πολλά ακόμα θα πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο ομάδας ή ομάδων. Η Άλτε πάντως προς το παρόν δεν μπορεί να παράσχει λεπτομέρειες. Βέβαια το θέμα είναι συλλογικό και θα επισώθουμε πάνω σε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Όπως και άλλες ομάδες, η Άλντε έχει κάποιες διαφωνίες, χρειάζεται χρόνος για να ασχοληθούμε με άλλα ζητήματα όπως η δημιουργία δεδομένων, η αρχή, η εργασιακή, η όλα αυτά που είναι τμήμα του πακέτου της κινητικότητας. Επιπλέον, το σύστημα αξιολόγηση κινδύνου για να δούμε ποιο είδος μεταφορών θα περιληφθεί σε αυτή την πρόταση. Λεπτό ζήτημα, αλλά βλέπει να υπάρχει ελπίδα. Παρ' όλα αυτά, μετά τη συνάντηση των σκιωδών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε σχέση με άλλα ζητήματα όπως το ρέο εργασία και τους επιτόπου ελέγχους, τεχνικές προσαρμογές και άλλα ζητήματα φαίνεται ότι η συζήτηση να πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Και θεωρεί ότι αυτές οι συναντήσεις των σχεδόν ήταν επικοδομητικές. Κατά την άποψη επίσης θα πρέπει να υπάρξουν συμβασμοί στις τροπολογίες για το χρόνο άπαυσης, το καποτάζ και θα πρέπει να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας. Πάντως δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα γίνουν όλα αυτά. Αν θα γίνουν δηλαδή σε επίπεδο εισηγητή ή αν θα εμπλακούν και οι σκιώδεις. Πάντως είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα θέματα είναι ελένδετα και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο σύνολο του φακέλου. Τέλος, χρειάζεται να διευκρινίσουμε τι γίνεται με την δήλωση απόσπασης. Οπότε η 191, 92, 193 94 ζητά να ληφθούν υπόψη από τον εισηγητή. Θα έλεγα κι άλλα, αλλά επειδή έχει περάσει ο... θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Merci, monsieur. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τελίνσκα. Εγώ παίρνω το λόγο τώρα γιατί είμαι συνεισηγήτρια σε αυτό το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, υπήρξε συμφωνία στην Επιτροπή Απασχόλησης επί της ε, Γενικής Οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων στους τριμερείς διαλόγους. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πραγματική νίκη για το σύνολο των εργαζομένων στην Ευρώπη, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, όποια και είναι το επάγγελμά του, ε, ε, ο χώρο δραστηριοποίησή του. Μιλούμε για ε, τους μισθούς, το 13ο μισθό και το καθεξής. Λοιπόν, πολύ καλή αυτή η συμφωνία στην Επιτροπή Επασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να είμαστε υπερήφανοι. Όμως, τίθεται το ζήτημα των μεταφορών. Διαβάζοντα ορισμένε τροπολογίε εδώ, δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει ειδική νομοθεσία στι οδικέ μεταφορέ που ξεφεύγει τελείω από το γενικό πλαίσιο τη οδηγία. Και κάποιε φορέ ε, αφαιρούνται ορισμένα δικαιώματα και έτσι πρόκειται για υποχώρηση σε σχέση με την γενική οδηγία. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα βεβαίω δεν λέω ότι θα πρέπει να είναι open bar η προσέγγιση, αλλά όπως και να έχει, αυτό αφορά μόνο τις οδικές μεταφορές. Και κάποιοι μπορούν να πούνε εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί μετακινούνται συνέχεια και δεν χρειάζεται να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Εγώ λέω όσο όχι πρέπει. Και θέλω να είμαι σαφής. Οι μεταφορές είναι ένας τομέας που πλήττεται από ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εξαιτία κοινότητα κινητικότητάς τους. Αυτή η οδηγή, και πολύ σωστά μας ανέφερε ο κ. Λούγκρεν που είναι και ο ίδιος οδηγός, ζη, ζουν ε, υπό απαράδεκτες ε, συνθήκες. Βλέπουμε την αγορά και διαπιστώνουμε σημαντικές διαφορές. Εγώ είμαι Ευρωπαία πολίτη, είμαι υπέρ τη ελεύθερη κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένα επαγγέλματα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί χρειάζονται κανόνες και αυτό το λέω γιατί αυτό το λέξη specialis δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να κάνουμε ε, τους οδηγούς ε, εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας στην Ευρώπη. Πρέπει οι κανόνες να είναι οι ίδιοι για όλους στην ενιαία αγορά. Στόχος εδώ δεν γίνεται να είναι να διατηρήσουμε την ε, ισορροπία ε, αγοράς ε, Υπονομεύοντα τα εργασιακά δικαιώματα. Επομένω, δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό το λέξη πεσιάλη έναν δούριο ύπο για να τροποποιήσουμε ε, τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, το ζήτημα τη ε, ε, της αποζημιωσής τους και το καθεξής. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει βάσει του άρθρου 91 που είναι και η νομική βάση ε, της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών πρέπει να κινηθούμε με διαφορετικό δρόμο. Από την άλλη δεν γίνεται να έχουμε ε, οδηγίες που στερούνται κάθε νοήματος. Πρέπει να μιλήσουμε για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Μόνο αυτό είναι το ζήτημα, το θέμα του ελέγχου. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε τα μάτια στο ζήτημα των ε, ε, ελαφρών εμπορικών οχημάτων. Γιατί σήμερα πρόκειται για μια πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι ο αριθμός του στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου έχει ε, εκτοξευθεί και αυτό τους επιτρέπει να ξεφεύγουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρέπει να δοθεί τέλος σε αυτό το φαινόμενο και όλα αυτά τα ζητήματα απαιτούν συγκεκριμένη απάντηση, γιατί στεκόμαστε στο χείλος του στο γκρεμού. Είτε θα βρούμε λύση, είτε δεν θα βρούμε το θάρρος να βρούμε λύσεις και εκεί δεν θα πρέπει να παραπονεθούμε όταν ε, θα έχουμε πέσει στον κρεμό, θα είναι πολύ αργά. Επομένως, πολύ απλό αυτό που θέλω να πω. Πρέπει να φέρουμε αποτελέσματα. Δεν γίνεται να υπονομεύσουμε τα δικαιώματα των οδηγών και ε, να υποβαθμίσουμε αυτή την κατηγορία εργαζομένων σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα πρέπει και οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών να βρισκόνται στο ίδιο επίπεδο. Αυτά ήθελα να πω, τα άπα και ησύχασα. Συνεχίζουμε. Όχι, γιατί πραγματικά νομίζω ότι σε αυτά τα προβλήματα δεν έχουμε περιθώριο σφάλματος. Πραγματικά. Κυρία Γιούτο δεν είναι εδώ. Η κυρία Λουκατσέσκα. Α, ο κύριος Λούνγκρεν πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. αρχικά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει, αλλά και την πρόεδρο Καρή Μαντέλη, γιατί πραγματικά έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι κάτι θα πρέπει να προσκομίσουμε εδώ ως αποτέλεσμα. Γιατί ορισμένες φωνές λένε εντάξει όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αστερική αγορά. Ναι εντάξει όντως. Όμως δεν είναι το δικαίωμα του καθενός να ε, πληρώνει μισθούς πείνας, ε, τους εργαζομένους με μισθούς πείνας και να τους ε, αναγκάζει σε συνθήκες σκλαβιάς να μένουν μέσα σε μια καμπίνα και να κοιμούνται εκεί. Χωρίς να φροντίζει τους κοινωνικούς δεσμούς και το καθεξής. βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με τα που είχαμε εντοπίσει το 2014 και αυτό καλό είναι. Προφανώς και υπάρχουν φορτηγά διεθνών επιχειρήσεων που θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα ε, να ε, κυκλοφορούν μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά, σαφώς, αλλά όχι σε βάρος των ε, δικαιωμάτων, γιατί τότε χάνουμε κάθε αξιοπιστία. Κάποια στοιχεία είναι θετικά η έλεγχη στο δικό δίκτυο. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μέσο που μπορεί να αξιοποιήσει η αστυνομία στα κράτη-μέλη για να διορθώσει τα κακό κείμενα. Και απαιτείται κάποιο μηχανισμό εδώ. Μια αρμοδιότητα που θα πρέπει να εκχωρηθεί στην αστυνομία. Ε, και σε όλο αυτό μπαίνει βέβαια και ο ευφύης ταχογράφος. Θα μπορεί λοιπόν η αστυνομία να δει πότε μπήκε, ε, πότε πέρασε τα σύνορα το φορτηγό, πόση ώρα, πόσες ώρες είναι και ο οδηγός, εγώ θα ήθελα οι ταχογράφοι να κατασταθούν πολύ νωρίτερα. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα. Όμω, θα πρέπει να δώσουμε ένα πραγματικό μέσο στην αστυνομία για να έχει εκείνη τα αποδεκτικά στοιχεία που απαιτούνται. Πρέπει να υπάρξει και απέτηση από τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι στα βαρέα φορτηγά. Γιατί υπάρχει τώρα αυτή η απέτηση, αλλά συχνά βλέπουμε ότι απλώς η αστυνομία μια συγκεκριμένη μέρα σταματάει ένα συγκεκριμένο αριθμό φορτηγών, βλέπει την άδεια και εντάξει, θεωρεί ότι έχει κάνει το καθήκον της. Αλλά πρέπει να έχουμε πραγματικούς σε βάθος ελέγχους από πραγματικούς ε, οδικούς επιθεωρητές που γνωρίζουν πώς λειτουργεί ένας τέτοιος ταχογράφος και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, θεωρώ. Όμως, με τα χαράς ακούω ότι όπως και να έχει βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ευχαριστώ, κυρία Λουκασέσκα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Από όλη αυτή τη συζήτηση σήμερα βλέπουμε ότι τώρα που έχει περάσει λίγο ο καιρός καταλαβαίνουμε ένα τον άλλον καλύτερα και αυτό είναι ε, μια θετική ένδειξη ότι θα καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Όμως μιλάτε συνέχεια για την εσωτερική αγορά, τις ελευθερίες και τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ Πιστεύω ότι αυτές οι αρχές είναι που θα ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος των εργασιών μας. Όμως, προσοχή, σε ό,τι αφορά την απόσπαση των εργαζομένων τώρα. Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται να συγκρίνουμε τους οδηγού με τους οικοδόμους, για παράδειγμα. Με έναν οικοδόμο που πάει στη Γαλλία για δυο τρει μήνες και παρέχει υπηρεσίε σε αυτή τη χώρα. Οι οδηγοί περνούν πολύ συχνά μόνο ε, φευγαλέα από μία χώρα ή περνάει μία μέρα στη μία χώρα, την επόμενη είναι σε άλλη. Επομένως, συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι η ε, διαμετακόμιση και το διεθνές εμπόριο δεν θα πρέπει να επαχθούν στην οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Σαφώς και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις απάτες και τις καταχρήσεις, όμως δεν ε, μπορούμε να αφήσουμε περιθώριο στις ε, ε, πλασματικές επιχειρήσεις όπου για παράδειγμα έχουν τον εργαζόμενο στη Γερμανία και παίρνει μισθούς Βουλγαρίας Ρουμανίας. Δεν συμφωνούμε με αυτό και κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Τώρα για τους ελέγχους. Είναι πολύ σημαντική, πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ χωρών. Όμως οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να οδηγούν σε υπερβολικό διοικητικό άχθος και κόστος, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσεις που δυσκολεύονται από αυτή την άποψη. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν οδηγό που να έχει μια στίβα χαρτιά δίπλα του. Θα πρέπει λοιπόν τα έγγραφα να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Τώρα για το καμποτάζ. Ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας Μιάνης ε, Νίλσεν. Ε, θα Έχουμε βέβαια και μία συνάντηση ε, των σχεδόν εισηγητών, όμως τα καμποτάζ ουσιαστικά από περιβαλλοντικής άποψης εισήχθη για το περιορισμό των εκπομπών διευθυντήτου άνθρακα. Και από αυτή την άποψη θα καταλήξουμε σε συμβιβασμό πόσες μέρες μπορεί να ισχύσει το καποτάζ. Γιατί δεν συμφωνώ με αυτούς που θέλουν να καταθέσουν τροπολογίες για να καταργήσουμε απολύτως το καμποτάζ. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα και να βρούμε τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό. Όμως όλοι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να το καταφέρουμε αυτό. Παρακαλώ κυρία Γαβούντα Ευχαριστώ. Συμφωνώ πολύ με τα όσα είπατε για τις ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, για την οδηγία ε, περί απόσπασης εργαζομένων, όπως και εσεί Και εγώ λυπάμαι που υπάρχει αυτή η κλαδική διάκριση σε βάρος των οδηγών. Βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε περαιτέρω το ισχύον δίκαιο. Η σχετική οδηγία ε, προβλέπει ε, Συγκεκριμένε διατάξει, οι οποίες γίνονται ε, σεβαστές. Τώρα νομίζω ότι η συγγήτρια και οι σκιώδη θα πρέπει να κάνουν μια διάκριση μεταξύ διεθνούς, ε, διεθνών μεταφορών και καμποτάζ. Η θέση μας για το καμποτάζ είναι σαφής και σε προηγούμενες ψηφοφορίες και οι κανόνες της απόσπασης ισχύουν από την πρώτη μέρα. Ναι, διαβάζει εξαιρετικά γρήγορα η ομιλήτρια φυσικά. Δεν υπάρχει έτσι και χρονική πίεση, οπότε πιο αργά. Ε, ακόμα και στην Επιτροπή Απασχόληση, ε, ακόμα και αυτοί που είναι υπέρ τη απελευθέρωση, αναγνωρίζουν αυτέ τι βάσει. Για τι διεθνεί μεταφορέ, αναγνωρίζω ότι η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, γιατί στην πράξη τη εφαρμογή τη οδηγία μπορεί να ε, οδηγήσει σε δυσκολίε. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την συγγήτρια τι θα έλεγε αν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες της χώρας στην οποία γίνεται η μετακόμιση Συγγνώμη που σας διέκοψε, λέει η Πρόεδρος, αλλά πραγματικά κανείς δεν καταλάβανε τίποτα. Κύριε Κόχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή Μέρια κύλων ευχαριστώ για την έκθεση. Θα είμαι σύντομος χρειαζόμαστε πρώτα αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και ταυτόχρονα δεύτερο μείωση του γραφειοκρατικού κόστους. Για παράδειγμα, να γίνεται στην έδρα της επιχείρησης ο έλεγχος των ωραρίων εργασίας και όχι σε ελέγχους καθοδών. Να αποτραπεί βέβαια οι χώρες μέλη να λάβουν προστατευτικά μέτρα με αυξημένη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, συμφωνώ να φύγουν ε, οι διαδρομέ transit, παρόλο που είναι σαφέ. ότι πρέπει ε, να, πρέπει να σημειώνεται αυτό διαρκώς. Από πότε θα ισχύει από ποιο ωράριο και μετά θα ισχύει ως ολόκληρη ημέρα, θα πρέπει να περάσει από τις 6 στις 9 ώρες αυτό. Ευχαριστώ πολύ και Κοχ. Κύριε Ρικέ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, διότι ήδη έχουν λεχθεί πολλά πράγματα και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι πράγματι θα κρίνουμε πιο πολύ προς το μέρος των εργαζόμενων, πιο πολύ προς το μέρος των επιχειρήσεων. Διότι υπερασπιζόμαστε τον τομέα των μεταφορών. Και όταν το κάνουμε αυτό φαίνεται μάλλον να υποστηρίζουμε τα δίκαια των επιχειρήσεων. Και εκεί υπάρχει διαφορά μεταξύ Ανατολή και Δύσης, με εξαίρεση στην Ισπανία. Όλοι βέβαια εδώ τόνισαν την ε, περιφερειακή διάσταση με έναν συναδελφό μας που έχει ήδη αποχωρήσει με επιχειρήματα τα οποία έχουν παραλυθεί πολλές φορές. Απόσπαση των εργαζομένων αποτελεί δόξα για την Ευρώπη κλπ. Παρόλο που κοινωνικά είναι τροπή. Έχουμε λοιπόν το στρατόπεδο το εθνικό, το ευρωπαϊκό, το στρατόπεδο των εργαζόμενων, των επιχειρήσεων κλπ. Όλα αυτά τα ακούσαμε σήμερα και δεν μιλούμε εδώ για φτωχού και πλούσιου όπω λέει η Νιέσα Αγιάλα Σέντερ. Τα έχουμε πει πάντω αυτά. Τώρα, η έκθεση τη κυρία Κίλονεν είναι ισορροπημένη. Βέβαια τώρα θα τραβήξουν η μένα από εδώ και από εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να φτάσουμε σε μια ακραία λύση που να διασπάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια πολύ μικρή πλειοψηφία υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης. Εγώ συμφωνώ με την Πρόεδρο ότι είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τον ευρωπαϊκό λαό ή τους ευρωπαϊκούς λαούς. Δεν μπορούμε να επιδεινώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζόμενων. Χρειάζεται πολύ μεγάλος προβληματισμός επ' αυτού. Δεύτερη παρατήρηση. Μπορούμε να υποστηρίξουμε την ιδέα ενός λέξη specialis, διότι οι εθνικέ και οι διεθνεί μεταφορέ δεν είναι μια οποιαδήποτε δραστηριότητα. Υπάρχει μια δυσκολία ανάμεσα στο να πάρουμε το γενικό πρόβλημα τη απόσπαση εργαζομένων και από την άλλη μεριά το ειδικό πρόβλημα τη απόσπαση οδηγών και να τραβήξουμε προ την την άλλη κατεύθυνση για να καταλήξουμε σε μια ακραία λύση. Χρειάζεται λοιπόν μια λύση ισορροπημένη που θα σεβαστεί ιδίω όμω το δικαίωμα των εργαζομένων. Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η απόσπαση των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα. Και διερωτώ με, μήπως προσπαθούμε εδώ να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Να ρωτήσω επίσης και να ζητήσω από την εισηγήτρια να ε, διατηρήσει την αρχή της ε, απλότητας. Είπατε και εισαγωγικά πολύ, ε, με πολύ στόμφο ότι το θέμα εδώ είναι το κοινωνικό dumping, αλλά νομίζω ότι ήσασταν πολύ αρνητικοί και δεν πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που στην πράξη να μην λειτουργεί. Από τη μία λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την Γενική Συμφωνία περί απόσπασης. Και εδώ μου κάνει εντύπωση ότι συνεχώς γίνεται λόγος για διαρθρωτική απόσπαση. Όταν λοιπόν κάποιος αποσπάται διαρθρωτικά, τότε θα πρέπει να προσαρμοστεί το εθνικό επίπεδο μισθού. Όμως στις μεταφορές συνεχώς έχουμε ε, διασυνοριακές μεταφορές και πολύ άνετα μπορεί ένα οδηγό φορτηγού να περάσει από τρει-τέσσερι χώρε μέσα σε μια εβδομάδα. Όλα αυτά κάποιο θα πρέπει να τα συντονίσει. Ε, ήδη από διοικητικέ άποψει υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και πολλή χαρτούρα και ξέρω ότι είναι επικίνδυνο το σχόλιο, αλλά πρέπει να προσέξουμε γιατί υπάρχει έλλειψη ε, οδηγών. 100.000 άτομα το 2025. Και δεν ε, μπορούμε να λύσουμε αυτή την έλλειψη με την απόσπαση. Θα το λύσουμε με καλύτερους μισθούς, οι οποίοι θα προκύψουν από την εσωτερική αγορά. Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό βέβαια με αυτό το 2025, αλλά το να βρούμε και να, συστήσουμε ένα, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα με τη τεράστια γραφειοκρατία που θα προκύπτει από την απόσπαση, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Έχω τις επιφυλάξεις μου. Τώρα, τι κάνουμε με τους μη Ευρωπαίους οδηγούς. Νομίζω ότι το είπε η κυρία Κιλόνεν. Όμως ε, βλέπουμε μια μεγάλη εισρωή οδηγών από Ουκρανία, Λευκορωσία, ακόμα και Τουρκία και Φιλιππίνες. που τους ε, έχουμε δει στα ευρωπαϊκά φορτηγά. Και αυτοί θα υπαχθούν στο καθεστώς απόσπασης. Ποιος το ελέγχει, ποιος το αποτρέπει. Θα ήθελα απλώς να το επισημάνω. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Wim van de Kamp, et je donne tout... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Van de Kamp. Η κυρία Βέρνερ, που θα μας προσφέρει την άποψη της Κομισιόν. Ναι, όταν μιλάμε για την απόσπαση των εργαζομένων, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπήρξε μια συμφωνία για τη σχετική οδηγία Μεγάλο βήμα δηλαδή πρόοδου. Η Κομισιόν ανέκαθεν έλεγε ότι ισχύει στο τομέα των μεταφορών όπως και σε άλλους τομείς. Όμως η πρότασή μας απέβλεπε στο να υπάρξουν συγκεκριμένε διατάξεις αναλογικές με την ε, πολύ με το πολύ κινητικό χαρακτήρα αυτού του τομέα, αυτού του κλάδου. Εδώ η κυρία Κιλόνεν θα πρέπει να με ότι ακριβώ θα πρέπει να βρούμε την σωστή δοσολογία των συστατικών για την επιτυχία. Για την ψηφιοποίηση τώρα, να πω δύο λόγια, του κλάδου του μεταφορών. Υπάρχουν ήδη αρκετά συστήματα. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε νέα για την ανταλλαγή δεδομένων και τους κανόνες εφαρμογής εδώ οι ηλεκτρονικοί κανόνες είναι, τα ηλεκτρονικά συστήματα ανταλλαγής είναι πολύ χρήσιμα, αλλά θα πρέπει να τα βελτιώσουμε, όχι να αυξήσουμε τον φόρτο. Και εμείς προσέχουμε ως Κομισιόν ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Για τις αποσπάσεις, νομίζω ότι έχουν προχωρήσει παντού οι συζητήσεις για το κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να ισχύει και η απόσπαση χρησιμοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις διατάξεις για τον κλάδο των μεταφορών. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι στις τροπολογίες προκύπτει διαφορά όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές και θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες διαφοροποίησεις όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της απόσπασης. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τις τροπολογίες θα σας, θα σας παρακαλέσω να έχετε υπόψη σας ότι χρειαζόμαστε απλούς κανόνες, ευκολονόητους και ευκολοεφάρμοστους. Και αυτό ήταν και το κινητρό μας όταν ε, προτείναμε συγκεκριμένο κατόφλι για άλλες τις διεθνείς μεταφορές. Και αυτό με οδηγεί στο να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τις διοικητικές προϋποθέσεις της εφαρμογής τον κανόνα για τις αποσπάσεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, περατός κατάλογος προϋποθέσεων ώστε να μην υπάρξουν διακρίσεις στην εφαρμογή και να υπάρχει και απαραίτητη ασφαλεία δικαίου για τους οδηγούς και για τις επιχειρήσεις. Επίσης η πρόταση της Κομισιόν αποβλέπει στο να αντιμετωπίσει προβλήματα που βλέπουμε σήμερα όπου οι διάφορες χώρες μέλη εφαρμόζουν διαφορετικές προποθέσει και αυτό δημιουργεί διοικητικό φόρτο. Θα πρέπει να πούμε ότι να έχουμε ένα ενιαίο, μια ενιαία δεσμή κανόνα από μόνη αποτελεί απλούστευση. Επίσης, βλέπουμε συμπαθητικά την ιδέα μόνο τα απαραίτητα έγγραφα διαθωρικούς ελέγχους να μεταφέρονται από τους οδηγούς έντυπα και ακόμα καλύτερα ηλεκτρονικά έγγραφα και ότι οι πληροφορίε είναι καλύτερο να ελέγχονται στην έδρα των επιχειρήσεων και όχι μόνο μέσω ελέγχων των οδηγών. Και αυτό αφορά βέβαια και το θέμα της αρχής ε, επιβολής. Τέλος, για τη διάκριση μεταξύ γενικών αποσπάσεων και επιμέρους κλαδικών αποσπάσεων για αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και άλλες διευκρινήσεις. Πάντως για την διαμετακόμιση θεωρούμε ότι αυτό δεν αφορά προσωρινή ή μακροχρόνια απόσπαση. Μάλιστα η μακροχρόνια απόσπαση αντιβαίνει στην ίδια τη φύση τη απόσπαση. Αυτό θέλω να το διευκρινίσω. Ευχαριστώ πολύ. Euh, ευχαριστώ κυρία Βέρνερ. Κυρία Κιλόνεν, για τη δευτερολογία σας. Παρακαλώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας Χαίρομαι που είμαι έτσι μια γυναίκα από το βορρά, δυναμική, με εξίσου δυναμικούς συνεργάτες, δουλευταράδες, μέρα νύχτα δουλεύουν για να βρούμε λύση. Υπάρχει και κάτι που θέλω να προσθέσω τώρα. Και θέλω να το σκεφτούμε. Κάθε φορά που αναφέρουμε εδώ το κοινωνικό ντάμπινγκ εδώ στο Κοινοβούλιο το τονίζουμε λες και να υπάρχουν εταιρείε που να δουλεύουν σωστά. Και επειδή εγώ προέρχομαι από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ξέρω ότι υπάρχουν πολύ καλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη που τηρούν την νομοθεσία που κάνουν ό,τι πρέπει και που προσέχουν τους εργαζόμενους τους. Δεν θέλω λοιπόν να τους τιμωρήσουμε όλους, γιατί δεν αφορά όλους αυτό το φαινόμενο. Επίσης, να καταλάβουμε ότι όταν αλλάζουμε την νομοθεσία, να λάβουμε υπόψη μας ότι χωρίς επιχειρήσεις δεν υπάρχει απασχόληση. Και είναι κάπως παράδοξο. Όταν αναζητούμε λύσεις λέμε ότι εντάξει θα τους τιμωρήσουμε όλους παρόλο που ξέρουμε ότι δεν εμπλέκονται όλοι. Το πρόβλημα είναι ότι αν αλλιώσουμε την αγορά και καταθέσουμε αυτή την πρόταση και προωθήσουμε το πρόβλημα στις τρίτες χώρες, τότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα στις μεταφορές στην Ευρώπη και αυτό δεν το επιθυμώ δεν θέλω να γίνει. Και νομίζω ότι φαίνεται ότι οι θέσεις μας σήμερα εξαρτώνται ή καθορίζονται από το αν καταγόμαστε από την Ανατολική ή Δυτική Ευρώπη. Καλό θα ήταν να αποφύγουμε αυτές τις διακρίσεις, αυτούς τους διαχωρισμούς. Και στο Συμβούλιο τρεις χώρες μέλη έχουν εφαρμόσει τους κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές. Γερμανία, Γαλλία και Αυστρία. Και να είμαι ειλικρινής ότι με αυτούς τους κανόνες που δεν σχεδιάστηκαν από τη σκοπιά των διεθνών αγορών και των μεταφορών, όλες αυτές οι υποθέσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και εγώ συμπονώ τους οδηγούς που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. και που εργάζονται η πλειοψηφία τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, αν για κάθε διέλευση συνόρων θα πρέπει να έχουμε έγγραφα απόσπαση, τότε θα επέλθει χάος. Και αυτό θα έχει επιπτώσει και στην απασχόληση των Ευρωπαίων οδηγών. Γιατί το πιθανότερο είναι να φύγουν δουλειέ και να πάνε σε τρίτε χώρε, όπω λέγαμε. Και δυστυχώ σε κάποιε περιπτώσει αυτό θα φορά και του αυτοαπασχολούμενους. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ κοινωνικών συνθήκων και ενιαίας αγοράς. Και, να το πω ξεκάθαρα, και προστατευτισμού. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να σκεφτούμε. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια ταυτόχρονα, αλλά νομίζω ότι επιγόντως χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα εμπιστοσύνη. Να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό. Να έχουμε δηλαδή μια πλατφόρμα όπου όλοι οι παράγοντες του εφοδιασμού θα μπορούσαν να αποδείξουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα και κανόνες. Οπότε αυτή η εμπιστοσύνη θα μπορούσε να δημιουργηθεί καλύπτοντας όλη την αλυσίδα των μεταφορών και ολόκληρο τον κλάδο γενικότερα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα επιβολής ή τιμωρίας, γιατί υπάρχουν και καλές εταιρείε, ξαναλέω, και καλοί επιχειρηματίε. Οπότε θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε αυτούς για να έχουμε μια πληρέστερη προσέγγιση, όχι, όχι μόνο τιμωρώντας τους παραβάτες. Τώρα για το θέμα της καμπίνας, της ανάπαυσης, της συνεχούς οδήγησης. Νομίζω ότι σας ήρθε κάτι ενημερωτικά. Ο, ο συνάδελφος εδώ πέρα, γι' αυτόν μιλάω, αλλά φαίνεται δεν με ακούει. Ναι, για σένα μιλούσα, αλλά δεν ακούγες, δεν ακούγες. θα πρέπει να μου στείλει φιλιά και λουλούδια και δεν ξέρω τι άλλο σε σχέση με τις αποσπάσεις. Γιατί θα βρούμε λύσεις. Πάντως είμαι σίγουρος θα βρεθεί λύση γιατί από τη στιγμή που είμαστε τόσο δεμένοι. Και συνεργαζόμαστε καλά. Ναι, αλλά μην φιλιώσαστε μόνο μεταξύ σα. Στείλε μου και κανένα και εμένα, λέει η ομιλήτρια. Τέλο πάντων, θα συνεχίσουμε τη δουλειά μα. Με συγχωρεί, Βίμ, δεν πήρα τα φάρμακά μου σήμερα το πρωί. Έτσι, οπότε γι' αυτό λέω αυτά που λέω. Αλλά σας παρακαλώ, καταλήγοντας. Αν έχετε κάποιες ιδέες να μου πείτε, έστω και αστείες και παράξενες, να μου τις στείλετε γιατί θα πρέπει εδώ να συλλέξουμε πραγματικά οποιαδήποτε δυνατή ιδέα για να σώσουμε τον κόσμο και τον πλανήτη. Έτσι. Ευχαριστώ. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιλονέν για αυτά τα λόγια αγάπης, λέει η Πρόεδρος. Βιν. Κλείνω την παρέθεση έτσι. Θα περάσουμε σε άλλα θέματα. Τροπολογίες. Να επιθυμίσω ότι στις 24 θα ψηφίσουμε, έτσι, 24 ώρα το πρωί, όπως και τις υπόλοιπες εκθέσεις. Πάντως, θα σας βοηθήσουμε κυρία Κιλονέν. Καλή επιτυχία και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το Ευρωκοινοβούλιο εγώ δυστυχώς θα πρέπει να φύγω γιατί έχω μια συνάντηση και για το τελευταίο θέμα για μια ώρα θα παραχωρήσω τη θέση μου στον κύριο Ρικέ. Αυτά ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στους διαδρόμους την επόμενη εβδομάδα στην Αλφή. Το θέμα αφορά τα μισθωμένα οχήματα στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ναι, με λύπη βλέπουμε να φεύγει η πρόεδρος μας, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει. Φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία μας έκθεση Πάμε λοιπόν στο θέμα αφορά την οδηγία χρήσης μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Η συγγήτρια κυρία Μοντέρο Δεαγκιάρ. Κυρία Μοντέρο Δεαγκιάρ, έχετε το λόγο. Σε δύο λεπτά θα έρθει η συγγήτρια. Μου είπαν. Δεν τη γλίτωσες. Τη γλίτωσες, λέει ο πρόεδρος. Yes. Voilà, si vous êtes euh, d'accord, et afin... Ωραία. Για να τελειώσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ την κυρία Μοντέρο που ήρθε και ζητώ το λόγο αμέσω για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της σε σχέση με τα μισθωμένα χήματα χωρίς οδηγό. Merci. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καστέρηση. Προσπαθούμε να λύσουμε παλιά προβλήματα, γι' αυτό άργησα. Για το θέμα αυτό, λοιπόν, που αφορά τι μεταφορές, καταρχάς να ευχαριστήσω του αδέλφους για τη συνεργασία τους, όπως επίσης και τη γραμματεία, που έκανε πολλά ώστε να εμβαθύνουμε σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι και αυτός ο φάκελος είναι αρκετά περίπλοκος, έχει τεχνικά ζητήματα και παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Και ιδιαίτερα αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι περιφερειακές που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες όμως καλύπτονται ή έχουν προσπάθεια να καλυφθούν στην έκθεση. Ο στόχος μας είναι εδώ, στην πρότασή μας, να έχουμε κάποια πρόνοια για τα οχήματα χωρίς που μισθώνονται. Και στοχεύουμε στο να υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι περιορισμοί, κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις και επίκλαμορφίες σε σχέση με αυτή την αγορά και ξέρουμε ότι υπάρχουν επίσης και διαφορές όσον αφορά τη ταξινόμηση σε εθνικό επίπεδο, χρονικές περίοδοι κλπ. Οπότε όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα λάβουμε υπόψη μας με τροποποιήσεις και με τροπολογίες όμως που κατατέθηκαν 81 συγκεκριμένα που θα προσπαθήσω να περιλάβω στην τελική μου πρόταση. Πάντως θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά που έχουν υποθεί επανειλημμένως σχετικά με διάφορες χώρες που όπου μάλλον είναι περισσότερο επιτακτικό να τροποποιηθεί η οδηγία. Όταν μιλάμε για αυτά τα οχήματα, μιλάμε για κάτι το οποίο έχει να κάνει με χρονικές ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, χρονική περίοδο της ε, μίσθωσης. Αυτό θέλουμε να το τονίσουμε στην πρότασή μας. Μάλιστα σήμερα το απόγευμα εδώ εμείς ε, συζητήσαμε κάποια θέματα που σχετίζονται άμεσα με αυτά εδώ. Και γι' αυτό και το λόγο θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μία νομοθεσία η οποία θα είναι ρεαλιστική, γιατί πολύ συχνά βέβαια μας κατηγορούν για το αντίθετο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού το βάρος το διοικητικό και σχετικά με τις αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να διευκολύνουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να διευκολύνουμε την σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις, απαντήσεις όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα στην οδηγία. Και τέλος θα ήθελα να πω το εξή για να μην με Θα ήθελα να πω και να τονίσω ότι εμείς κατανοούμε και, προσ... και προσδίδουμε τη δέουσα σημασία στο θέμα της ε, προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να προσπίσουμε τις συνθήκες εργασίας αυτών των εργαζομένων αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάποιους διαχωρισμούς. γίνεται λόγος για εκπαίδευση, κατάρτιση, διαβίου μάθηση των οδηγών. Οδηγία 2389. Οπότε βεβαίως θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας την ε, κατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την προάσπιση των εργαζομένων, αλλά εδώ και πάλι ξαναλέω δουλεύουμε πάνω σε ένα κείμενο το οποίο αφορά οχήματα χωρίς οδηγό για εμπορευματικές μεταφορές, οδικές. Αυτά είχα εγώ να σας πω, προκατακτικά. Ήδη έχουμε την πρώτη συνάντηση των σκιωδών και προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε και να διερευνήσουμε τις κόκκινες γραμμές της κάθε πολιτικής ομάδας. Προσπάθησαμε πάντως να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της αγοράς. Προσπαθώντας βέβαια να μην δημιουργήσουμε νέους ε, φραγμούς, να μην δημιουργήσουμε μέτρα ή υπερβολικά δεσμευτικά, ώστε να έχουμε τελικά ένα έγγραφο τελικό που θα είναι ισορροπημένο και γι' αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω να δεχτώ να αποδεχτώ όσες περισσότερες τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Άντερσον, σκιώδη συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και το επιτελείο της για την πολύ προσεκτική δουλειά που έχουν κάνει σε αυτό το φάκελο και για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει μέχρι τώρα. Ήταν εξαιρετικό το σεμινάριο που διοργανώσαμε από κινούμε μία σειρά φορεί. Να ευχαριστήσω για τη γραμματεία, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η προσέγγιση αυτό το φάκελο. Συμφωνούμε σε μεγάλο αριθμό θεμάτων. Είναι σημαντικό το ζήτημα. Θα πρέπει να το εξετάσουμε για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί σωστά η αγορά ε, με έναν ε, σωστά διευθετημένο τρόπο. Να υπάρχει λοιπόν σωστό κανονιστικό πλαίσιο. Παρά το δεν υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για αυτό το φάκελο, εμεί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Υπάρχουν ζητήματα όπω ε, η επιβολή του νόμου, ότι τα μισθωμένα οχήματα δεν θα επανομεύουν όλα όσα εξετάζουμε εν γέννη σε άλλου τομεί από πλευρά επιβολή του νόμου. Ζητήματα όπω η βάση δεδομένων, η καταχώρηση, οι πινακίδε και πολλά άλλα ζητήματα που άπτονται τη ασφάλεια και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των μισθωμένων οχημάτων. Και να είμαι σαφή εδώ σε ό,τι αφορά στην αναφορά που κάνατε στους σοσιαλδημοκράτες, ούτε εμείς ούτε κανένας άλλος δεν μπορεί, ε, δεν προσπαθεί να βάλει εργατικά δικαιώματα κάτι άλλο εδώ. Απλώς όταν υπάρχει σωστή κατάρτιση ε, για να έχουμε ευρύτερη κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου, αυτό αυξάνει την ασφάλεια αποφεύγουμε έτσι προβλήματα και ένα από αυτό που ανέφερε η Επιτροπή για τα μισθωμένα οχήματα είναι ότι ακόμα και από περιβαλλοντική άποψη είναι πιο αποτελεσματικό να έχουμε πιο καινούρια μισθωμένα οχήματα. Βέβαια, δεν θέλουμε να, να ρυθμίσουμε το πλαίσιο των οδηγών απαραίτητα, απλώ να διασφαλίσουμε ότι θα είναι σε θέση να οδηγήσουν αυτά τα οχήματα με τον κατάλληλο τρόπο για να μεγιστοποιήσουμε και τα ωφέλη. Οπότε εδώ δεν πρόκειται για εργασιακά δικαιώματα ή κάτι άλλο. Θέλουμε ένα γενικό πλαίσιο που να ε, ωφελήσει εν γέννη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Άντερσον. Εξ ονόματος ε, του ECR νομίζω δεν υπάρχει κανείς. Για την άλλη ο κύριος Τέλιτσκα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς είναι απόν ο σκιώδης μας κύριος Μίλτενμπεργκ διότι έχει άλλη ανηλυμένη υποχρέωση, με παρακάλεσε να μιλήσω εγώ εκ μέρους του και να τονίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτα, να αφαιρέσουμε τις περιστε... τους περιτούς περιορισμούς και να επιτρέψουμε να λειτουργήσουν ε, οι επιχειρήσεις αυτές όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται ωστόσο κάποια μίνιμουμ ρύθμιση. Οι περιορισμοί θα πρέπει να είναι αναλογικοί. Πρώτα, οι χώρες μέλη θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν αυστηρότερη την... Ε, ε βάζουν ευθυρότερους περιορισμού, 25% μόνο του στόλου. Όταν ο στόλος είναι λιγότερο από τέσσερα αυτοκίνητα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται ένα από αυτά. Οι χώρες μέλη θα επιτρέπουν την χρήση υβριδικών αυτοκινήτων για τέσσερους συνεχείς μήνες για να αντιμετωπίζονται οι κορυφώσεις στην αγορά. Οι χώρες μέλη επίσης, με συγχωρείτε, δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πλέον να περιορίζουν τη χρήση υβριδικών οχημάτων κάτω των 6 τόνων για διάφορες, ε, για διάφορες ε, επιχειρήσεις. Τροπολογίες θα υποβληθούν για, την, ε, για τον περιορισμό, για την διατύπωση μάλλον αυτών των περιορισμών. Ευχαριστώ. Α, με συγχωρείτε, η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Η Νέση, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, πρόεδρε όχι για, τα, για τις μεταφορές αλλά για τα μισθωμένα οχήματα γενικότερα. Να πω προς την Κομισιόν το εξή. Υπάρχει η δυνατότητα σχετικά άμεσα να θεσπίσουμε νομοθεσία για την μίσθωση οχημάτων ώστε οι επιχειρήσεις να κάνουν εναρμονήσεις επειδή το να μισθώσει να μισθώσει κανείς ε, ένα όχημα σε μια πόλη και να το παραδώσει σε άλλη πόλη εντός της χώρας εντάξει αυτό συμβαίνει αν όμως γίνει από μια χώρα στην άλλη όπως συνέβη σε μένα βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο Οπότε μήπως σε κάποιο σχετικά άμεσο μέλλον θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ένα πλαίσιο εναρμόνισης για τα έθη και τα έθιμα της μίστοσης, η ώστε να μην μας βγαίνει ο κούκος και να μπορούμε να μισθώνουμε ανεξέλεκτα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς κυρία Βέρνερ είστε ακόμη εδώ. Μάλιστα. Έχετε το λόγο πάλι ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια κυρία Μοντέρο και τους ε, διάφορους ευρωβουλευτές για τις παρεμβάσεις τους. Δεν πρόκειται για κοινωνικού χαρακτήρα πρόταση. Πρόκειται για κλασική πρόταση ενιαίας αγοράς. Έχουμε αριθμό χωρών μελών που επιτρέπουν ήδη στους επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα και σε άλλες χώρες μέλη και κανείς από αυτούς δεν επισημαίνει σημαντικά προβλήματα. Εμείς βλέπουμε κάποιες δυνατότητες αύξησης της αποτελεσματικότητας, άρση περιορισμών που θα επιτρέψουν στους επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν ε, τις περιόδους ε, κορύφωσης των εργασιών. Και η βασική αρχή στο άρθρο 2 της προτάσεως λέει ότι όταν ένας επιχειρηματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει μισθωμένο όχημα στην χώρα του, στη χώρα της έδρας του δηλαδή, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως του που είναι ταξινομημένο το όχημα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί κάποια χώρα μέλος άλλη εκτός από την έδρα να έχει τη δυνατότητα να επαγορεύει τους κανόνες. Υπάρχουν όμως και κάποιοι και κάποιες τροπολογίες για το άρθρο 2 που εμείς θεωρούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μάλλον ταιριάζουν στο άρθρο 3 το οποίο άρθρο 3 επιτρέπει στην χώρα της εγκατάστασης να προβλέψει κάποιους περιορισμούς και ορισμένοι από τους περιορισμούς αυτούς προερχόνται από την επιθυμία των χωρών να αποτρέψουν την φοροαποφυγή. Βεβαίω η φορολογία των οχημάτων ποικίλει από μια χώρα μέλο σε άλλη. Άρα υπάρχει πράγματι η δυνατότητα οι επιχειρηματίε να ταξινομούν τα οχήματα σε άλλε πιο ενδιαφέρουσε δικαιοδοσίε, και αυτό ίσω επιθυμεί η χώρα μέλο τη εγκατάσταση να το αποφύγει. Στην πρότασή μα. περιλαμβάνουμε ένα τέτοιο περιορισμό για να το αποφύγουμε αυτό, περιορίζοντα δηλαδή την διάρκεια χρήσης του μισθωμένου οχήματος. Ορισμένες τροπολογίες στοχεύουν στην μείωση αυτής της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης σε ένα μήνα. Όμως αυτό είναι υπερβολικά δραστικό μέτρο και έρχεται αντίθετο στην ανάγκη αντιμετώπισης ε, των ε, κορυφώσεων της απασχόλησης ε, δραστηριότητας. Τροπολογίες που επιτρέπουν στις χώρες μέλη να συνεχίσουν να περιορίζουν τη χρήση των μισθωμένων οχημάτων για επιχειρήσεις για τον ίδιο λογαριασμό τους, αυτό είναι αντίθετο με την αρχική πρόθεση της Κομισιόν. Όπως είπα, τα μισθωμένα οχήματα μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και ευκαμψία των επιχειρηματιών και δεν βλέπουμε λόγο για τον οποίο να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τις ε, επιχειρήσεις που γίνονται, τις ε, ενέργειες δηλαδή που γίνονται για τον ίδιο λογαριασμό. Εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει άλλη επιλογή, μπορεί να αγοράσει όχημα και να το υποχρησιμοποιεί. Και γνωρίζουμε ήδη ότι κατά μέσον όρο αυτό θα οδηγήσει σε ε, στόλους οχημάτων μεγαλύτερης ηλικίας. Κατά μέσον όρο υψηλότερης ηλικίας σε χώρες με περιορισμούς από αυτές που είναι σε χώρες χωρίς περιορισμούς. Και μία από τις κοινέ κόκκινες γραμμές σε όλες τις προτάσεις είναι για την επιβολή. Η επιβολή θα πρέπει να γίνεται με χαμηλό κόστος και χαμηλή γραφειοκρατική επιβάρυνση και γι' αυτό υποστηρίζουμε τις τροπολογίες εκείνες που αναφέρονται στη χρήση ψηφιακών μέσων και ιδίω των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για όλες τις επιχειρήσεις μεταφορών. Η, δε πινακίδα του κάθε οχήματο θα πρέπει να είναι να καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο στο εθνικό μητρό και εξετάζοντα το μητρό αυτό, οι αρχές θα πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν ποιο όχημα είναι ίδια ιδιοκτησία του επιχειρηματία και ποιο είναι μισθωμένο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη, δηλαδή την αναλογικότητα των μέσων και υπό αυτό το πρίσμα θα θέλαμε να εξετάσετε και εσείς τη συγκεκριμένη τροπολογία. Συνολικά, η πρόταση αυτή θα βοηθήσει τους επιχειρηματίες, θα κάνει πιο αποτελεσματική την ενιαία αγορά, θα άρει κάποιους από τους κανόνες που οικονομικά δύσκολα μπορούν να αιτιολογηθούν. Στην ουσία πρόκειται περί της αναλογικότητας των ρυθμίσεων, που θέλουμε, όπως είπα, η ρύθμιση να είναι αναλογική. Σας ευχαριστώ, κυρία Βέρνερ. Εν τέλει, η εισηγήτρια ε, να πει τα τελευταία λόγια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να πω το εξής. Στην τελευταία συνάντηση των σκιωδών είχαμε συμφωνήσει ότι θα λάβουμε υπόψη τα άρθρα 2 και 3 τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν χωριστά. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συζητήσουμε αφενός και να λάβουμε υπόψη αφενός το κόνσεπτ αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις, ιδίως την κυρία Γιάλα Σέντερ, που δεν ήταν άμεση η σχέση βέβαια με το υπεριεχόμενο της εκθεσής μου, σχέση του σχολείου δηλαδή, αλλά είχε πάντως κάποια σχέση με μισθωμένα οχήματα ο πρόεδρος, ο προεδρεύων Ρικέρ. Η ψηφοφορία θα εξαχθεί όπως και τους άλλους φακέτους κινητικότητας στις 24 Πέμπτου και ε, από τις 9 το πρωί, αλλά νομίζω ότι θα διαρκέσει και όλο το πρωινό. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις στην φάση αυτή της ε, συναντήσεώς μας. Θεωρώ ότι λίγη εδώ. Το επόμενο ραντεβού μας είναι στις 12 Απριλίου 9 το πρωί. Πέμπτη λοιπόν 9 το πρωί. Ευχαριστώ και καλό σας απόγευμα.